Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από ένα εκπρόσωπο τη κυρκασική αντιπροσωπεία να λάβει το λόγο για να γνωρίζουμε ότι υπάρχει τέτοιο λαό και ότι υπάρχει μια τέτοια κατάσταση στο Βόρειο Κάφκασο και στον κόσμο. Σα παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ια Ντιουάρ, είμαι Κυρκάσιος. Ο λαός μου λέγεται Κυρκασί. Η πατρίδα μας είναι η Κυρκασία στο βορειοδυτικό Κάφκασο. Από το τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα αντιμετωπίσανε οι συμπολίτες μου, ο λαός μου, δράσεις γενοκτονίας που οδήγησαν στην αναγκαστική εκτόπιση 1,2 εκατομμύριων ανθρώπων. Ο συνολικός πληθυσμός είναι περίπου 2,5, ήταν τότε 2,5 εκατομμύρια, 60% εσφάγησαν ή πέθαναν από το λοιμό ή διασκορπίστηκαν στο μεγαλύτερο μέρος του όλου του κόσμου, έχουν μεγαλύτερη διασπορά. 90% από εμά είναι εκτός Καυκάσου και μόνο 10% είναι στον Κάυκασο Και μέσα και έξω από τον Κάυκασο εξακολουθούμε να υφιστάμεθα τις συνέπειες της γενοκτονίας που διεπράχθηναν δύο του λαού μας που έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα στην χώρα μας, στο Βόρειο Κάφκασο, λαμβάνουν χώρα πολλές ε, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θέλουμε ο κόσμος και η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει κάποια προσοχή ώστε να μπορέσουμε να καταπραίνουμε τα θέματα αυτά. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες που θα γίνουν στην, προστα... στην ε, πρωτεύουσα της πρώην Κυρκασίας του Σότσι, χειμερινή Ολυμπιακή, το Σότσι ήταν και ο χώρος όπου έγινε μια μεγάλη γενοκτονία των κυρκασίων στο παρελθόν και τα σχέδια της δημιουργίας εγκαταστάσεων για τους Ολυμπιακούς του 2014 στο Σότσι δημιουργούν μεγάλα προβλήματα και αγωνία στο λαό μας και μέσα και έξω από, τον, από την Κυρκασία. Πρόκειται για βλάβη στο περιβάλλον τη συνέπειες αυτής της κατασκευής που θα έχει επιρροή σε όλη την περιοχή και θα επηρεάσει το μέλλον του λαού μας. Πέραν της διαφθοράς και των καταχρήσεων σε επίπεδο κυβέρνησης έναντι του λαού, έναντι των οικονομικών πόρων και έναντι της έγκυας περιουσίας για τη δημιουργία του συμπλέγματος στο Σότσι, το σχέδιο του Ολυμπιακών του Σάτσι είναι σε παραβίαση των κανόνων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής που, απαγορεύουν τη χρήση χώρων όπου έχει διαπραχθεί γενοκτονία. Ζητούμε λοιπόν από τους λαούς όλου του κόσμου να κατανοήσουν την τραγωδία μας, τη γενοκτονία που υπέστημε, την πραγματικότητα του Καυκάσου και όλα, όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Καύκασο και τη βλάβη στο περιβάλλον. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που μας δίνετε να λάβουμε το λόγο σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την ευκαιρία να είμαστε εδώ. Um, Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρο. Θα πρέπει πράγματι να δώσουμε σημασία στα προβλήματα αυτά τα οποία προκύπτουν από τη δημιουργία του Ολυμπιακού Συμπλέγματο στο Σότσι. Πολλοί μου έχουν αναφέρει οι και άλλοι που θεωρούν ότι υπάρχει παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών σε αυτή τη διαδικασία και δεύτερον θέλω να πω Ό,τι κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βόρειο Κάφκασο είναι πάντα στο επίκεντρο τη προσοχή μα. Γνωρίζουμε πόσο οδυνηρή είναι η κατάσταση εκεί. Ξέρουμε ότι είναι πραγματικά πολύ δυσμενή τα πράγματα. Τρει από εμά ήταν μέρη μια αντιπροσωπεία στη Βόρεια Οσετία και την Ιγκουσιατία πριν από μερικέ εβδομάδε. Μπορέσαμε να συναντήσουμε με οικογένειε ατόμων που είχαν ε, απαχθεί, βασανιστεί ή απλώς εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει τέρμα στο, στους βασάνους του λαού εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ θα αντιμετωπίσουμε αργότερα φέτος το θέμα αυτό. Και τώρα θα ήθελα, θα ήθελα να σταθώ στην απογευματινή μας ακρόαση που αφορά τη μεγάλη ανάγκη αντιμετώπιση τη ατιμορρησία, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για όλο τον κόσμο. Έχουμε το παράδειγμα τη Αργεντινή, όπου ε, εμπλέκεται και η υποεπιτροπή μας. Είναι απαραίτητο να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε την ατιμορρησία σε παγκόσμιο επίπεδο και να φέρουμε τους υπευθύνους ενώπιον της διεθνούς δικαιοσύνης. Έχω την, ε, είχα την ευκαιρία να συναντηθώ την Τρίτη με τον, <clears throat> με τον κύριο Άλμπερ Γκαλότο, τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της Αργεντινής και με ενθάρρυνε ιδιαίτερα η στάση του σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τη χώρα του την Αργεντινή για να αντιμετωπιστεί το οδυνηρό παρελθόν της δικτατορίας στην Αργεντινή για το οποίο θα ακούσουμε περισσότερα σήμερα το απόγευμα. Έχουμε τρεις διακεκριμένους ομιλητές σήμερα τον δόκτορα Δανίλ Εδουάρδο Ραφέκας, ο οποίος ποδιακός δικαστής στην Αργεντινή καταρχήν. Στη συνέχεια τον Ροδόλφο Γιανθών, ο οποίος είναι δικηγόρος αγωνιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρόεδρος της Ένωσης του ιδρύματο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τη Αργεντινή και ο τρίτο διακεκριμένο ομιλητή μα είναι ο κύριο Ρέμες Λένισοφ, τη Αργεντινή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως θα μιλήσει λίγο πιο σύντομα από τους προηγούμενους δύο ομιλητές. Και φυσικά θα ακούσουμε και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα αυτά. Θα μπορούσα λοιπόν να προσκαλέσω τον δόκτωρα Ραφέκας για να λάβει το λόγο παρακαλώ να μας εξηγήσει την κατάσταση του πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ομότητες και τις βιαιότητες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της πρώην δικτατορίας που υπήρχε στην Αργεντινή πριν από μερικά χρόνια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί για μένα είναι μια πραγματική τιμή να εκπροσωπήσω εδώ την Αργεντινή και τη δικαιοσύνη της Αργεντινής. Πράγματι, μεταξύ του 1976 και του 1983 στην Αργεντινή υπέστη με τις συνέπειες μιας οδυνηρής και αιματηρής δικτατορίας, στρατιωτικής δικτατορίας. 30.000 άτομα ήταν κρατούμενοι, πολλοί από αυτούς εξαφανίστηκαν, ήταν αγνοούμενοι. Μισό εκατομμύριο Αργεντινοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, να πάνε σε άλλες περιοχές της χώρας από τις αιστείες τους ή ακόμα και να φύγουν στο εξωτερικό. Αυτός ο απολογισμός λοιπόν ο ιδιαίτερα ζωφερός συνοδεύεται με την ε, στάση του αυταρχικού καθεστώτος στην Αργεντινή που θέλησε να προχωρήσει σε μια ουσιαστική πολιτιστική αλλαγή της αργεντινής κοινωνίας θέλοντας να τη μετατρέψουν σε ένα κάθετο αυταρχικό αντιδημοκρατικό καθεστώς. Τα τελευταία πέντε χρόνια περίπου η Αργεντινή για πρώτη φορά στην ιστορία της προβαίνει σε μια προσπάθεια να δει με καθαρά μάτια το πρόσφατο παρελθόν της, αυτό με μια κρατική πολιτική που περιλαμβάνει και τους τρεις πυλώνες του σύγχρονου δημοκρατικού κράτους Αργεντινής και έχει σαν κύριο άξονα τη δικαστική εξουσία, το ανώτατο δικαστήριο και τα δικαστήρια από τα οποία προέρχομαι και εγώ και μετά από τη μεγάλη αποτυχία πολιτικών που επί 25 χρόνια προσπάθησαν να οδηγήσουν στην αμνηστία, στην λύθη, στην ατιμορρησία και υποτιθέμενη συμφιλίωση μεταξύ των Αργεντινών. Όλες αυτές οι πολιτικές κατά την άποψή μας δεν οδήγησαν πραγματικά πουθενά. Ήταν μια απώλεια χρόνου. Τα τελευταία όμως πέντε χρόνια έχουμε ξεκινήσει να ακολουθούμε ένα δρόμο ο οποίος φαίνεται πια ότι είναι ο σωστός δρόμος, ο δρόμος της ανάμνησης, της μνήμης, της αποκάλυψης της αλήθειας, της δικαιοσύνης. Και όταν αναφέρομαι σε, δικαιοσύνη μιλάω για δίκη και κυρώσεις για όλους τους υπεύθυνους από τα υψηλότερα επίπεδα μέχρι τους βασανιστές, βιαστές και απαγωγείς Από αστικά, από πολιτικά δικαστήρια, στα ίδια πολιτικά δικαστήρια στα οποία κολλάζονται οι δράσεις οποιοδήποτε αδικοπράτοντας και μέσα στα πλαίσια των εγγυήσεων των δικονομικών όλου του δικαστικού συστήματος Αργεντινής. Και πάντα βασιζόμενοι στις, στην ποινική νομοθεσία που ήταν εν ενεργεία τη στιγμή που διαπράχθησαν τα εν λόγω αδικήματα. Πρόκειται λοιπόν κάτι το οποίο εμεί προσπαθούμε να φέρουμε σε πέρας τα τελευταία πέντε χρόνια πιστεύω ότι το κάνουμε με τρόπο επιτυχημένο. Είναι μια διαδικασία δικαστική δίωξη των υπευθύνων όλων αυτών των εγκλημάτων της δικτατορίας και θέλουμε με τον τρόπο αυτό να καταδείξουμε και την ηθική υπεροχή της δικαιοσύνης μιας δημοκρατίας, τη δικαιοσύνης ενό κράτου δικαίου έναντι αυτού που υπήρξε μια αστυνομικού χαρακτήρα δικαιοσύνη η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης δικτατορίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου χίλια άτομα τα οποία είναι κατηγορούμενοι στις διάφορες δίκες. Πολλοί από αυτούς έχουν ήδη καταδικαστεί αυτή τη στιγμή στην Αργεντινή λοιπόν προχωρούν δεκάδες από δίκες εναντίον αυτών των ε, κατηγορουμένων σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Αργεντινής και αυτές οι δίκες μέσα από τα μέσα ενημέρωσης αντανακλούν και κάνουν δημόσιες τις ιστορίες, τις δικατορίες, τις δολοφονίες, τις απαγωγές παιδιών, τους, ε, τις απαγωγές των θυμάτων και με αυτόν τον τρόπο, μετά από 30 χρόνια, επιτέλους, μετά από 30 χρόνια λύθης και ατιμορροσίας, καταφέρουμε να σπάσουμε τον τείχο της σιωπής, το τείχος της ατιμορρησίας που είχε με μεγάλη προσπάθεια δημιουργήσει η δικτατορία στην Αργεντινή και η συνενοχή της. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια χρονική στιγμή στην οποία η κοινή γνώμη και η κοινωνία της Αργεντινής μπορούν επιτέλους να λάβουν γνώση των ακροτήτων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της δικτατορία του κρατικού, της κρατικής τρομοκρατίας της δικτατορίας και αυτή η γνώση της ιστορικής αλήθειας είναι κάτι το οποίο οδηγεί σε μια αυξανόμενη αλληλεγγύη, αυξανόμενη υποστήριξη, αυξανόμενη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών για άλλες αυτές τις διαδικασίες που οδηγούν στη συλλογική μας μνήμη, στην απόδοση δικαιοσύνη έναντι αυτής της πολιτικής του δικτατορικού κράτους στην Αργεντινή. Όλα αυτά χωρίς όχι οδύνη, χωρίς βάσανα, χωρίς μια οδυνηρή ανάμνηση. Γιατί η τίμια αυτή αναζήτηση και ανάπλαση του παρελθόντος είναι ιδιαίτερα οδυνηρή και, να μας, και μας οδηγεί να κατανοούμε ότι είναι ίσως η πιο μαύρη ιστορία της ιστορίας της Αργεντινής σαν χώρας. Αυτά τα οποία έλαβαν χώρα την εποχή της δεκτατορίας. Την εποχή αυτή που υπήρξαν 300 παράνομα και κρυφά κέντρα ε, κράτησης βασανιστήριων και υποχρεωτικής εξαφάνισης κέντρα όπου είχαν πολλά στοιχεία κέντρων συγκέντρωσης όπου τα θύματα αυτών των κέντρων υφίστανται μια διαδικασία απανθρωπισμού. Μια βία διαδικασία απανθρωπισμού. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν που έφερε τον Ροδόλφο Σανσόν και μένα από το Buenos Aires ως εδώ μπροστά σας, στην Επιτροπή σας, μέσα στα πλαίσια λοιπόν αυτής της πολιτικής η οποία λαμβάνει η χώρα σήμερα στην Αργεντινή, εμείς ως πολίτες της Αργεντινής διαδραματίζουμε ένα ρόλο ο οποίος είναι ένα στίχημα σε σχέση με το μέλλον και το παρόν της χώρας μας. Γιατί για πρώτη φορά αρχίζουμε οριστικά να απομακρυνόμαστε από μια αυταρχική κουλτούρα. Μια κουλτούρα η οποία το, με τη φωτιά και το τσεκούρι επιβλήθηκε από τους δικτάτορες της Αργεντινής. Μέσω αυτών των διαδικασιών πραγματικής ανάμνησης, μνήμης, συλλογική και δικαιοσύνης που προξενεί σε όλους μας μια συλλογική μεγάλη οδύνη, μπορούμε επιτέλους σε ουσιαστικό επίπεδο να εδραιώσουμε το δημοκρατικό σύστημα στη χώρα μας το οποίο επισήμως τυπικά ίσχυε από το 1983, αλλά μόνο τα τελευταία χρόνια πραγματικά ριζώνεται και εδρεώνεται σε βάθος στην Αργεντινή μας. Με το να απομακρυνόμαστε οριστικά, και το τονίζω αυτό, από την αυταρχική αυτή κουλτούρα που σώβησε στη χώρα μου σε ένα μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα που σημαδεύτηκε από επανειλημμένα πραξικοπήματα και περιόδους στρατιωτικής δικτατορίας. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα το οποίο ήθελα να συμμεριστώ μαζί σας με εσά ως εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε σχέση με την μεγάλη σημασία που επέχουν αυτές οι διαδικασίες για το παρόν και για το μέλλον της Αργεντινής σας χώρας και επίσης πιστεύω ότι δεν χωρεί καμία αμφιβολία ότι με ένα έμεσο τρόπο αυτή η διαδικασία έχει επιπτώσει και σε όλες τις άλλες χώρες της περιοχής μας όπου υπήρξαν και εκεί στρατιωτικές δικτατορίες και αναπτύχθηκαν διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης του παρελθόντος στις αδελφές χώρες μας, στη Λατινική Αμερική. Και οίκοθε εννοείται ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει έμφαση, να υπογραμμίσει τη σημασία αυτών των διαδικασιών που περνάνε μέσα από θεσμικούς διάβλους, μέσα από διαφορετικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορέσει να γίνει σαφές με τρόπο επίσημο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει αυτή τη διαδικασία αντιμετώπισης του παρελθόντος γιατί δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ξεχάσουμε ότι και στην Αργεντινή έχουμε να αντιμετωπίσουμε αντιπάλους οι οποίοι είναι στη μειοψηφία προς το παρόν αλλά οι οποίοι προσπαθούν να αλλοιώσουν αυτή τη διαδικασία και να την υπονομεύσουν. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ε, δυνατότητα να λάβω το λόγο σε εσά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα καλά νέα αυτά που μας ε, φέρνετε από την Αργεντινή κύριε Ραφέκα. Συνήθως δεν ακούμε καλά μαντάτα. Ε, αντιμετωπίζουμε σοβαρές και συνεχιζόμενες παραβιάσεις ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που θα λάβει η χώρα μετά, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και πώς ε, η εμπειρία της Αργεντινίας μπορεί να βοηθήσει την καταπολέμηση της ατιμορρησίας σε άλλα μέρη και τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη, για να διδαχτούμε τα μαθήματα που πρέπει. Σήμερα το πρωί κάναμε μια σοβαρότατη συζήτηση για την κατάσταση στην ε, Βυρμανία, κάθετος Μιανμάρ, και μια και η Αργεντινή είναι ενεργό μέλος του Διεθνούς Μηχανισμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα να ακούσω από εσά τι ιδέες έχετε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Βυρμανίας όπου ο λαό τη χυμάζεται ε, από ένα σκληρό καθεστώ. Αλλά πρέπει να περιμένουμε γιατί έχουμε να ακούσουμε τώρα έναν επόμενο μιλητή, ε, δικηγόρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον κύριο Γιάνσον. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όπως και ο κύριος Ραφέκας για την ευκαιρία που μας δίνετε να λαμβάνουμε το λόγο ενώπιόν σας στην Επιτροπή. Διάβαζα με προσοχή την έκθεση που έχουν όλοι οι σημερινοί παρευρισκόμενοι όπου περιγράφεται η κατάσταση της καταπολέμησης της ατιμορρησίας στην Αργεντινή και η έκθεση αυτή τονίζει ένα θέμα που είναι πολύ ανησυχητικό Και είναι εξή κατάσταση. Εδώ και τέσσερα χρόνια παραμένει κάποιος αγνοούμενος, ο Χόρχε Χούλιο Λόπες, που ήταν επιζών μάρτυρας της δικτατορίας και πριν από τέσσερα ε, χρόνια ε, κατέθεσε ως μάρτυρα σε μια δίκη και έκτοτε εξαφανίστηκε. Και μέχρι σήμερα δεν έχουμε κανένα νέο του. Αγνοείται πλήρως και θα πρέπει να συνεχίζουμε να το διατρανώνουμε αυτό και να το λέγουμε παντού όπου έχουμε την ευκαιρία και στο εσωτερικό αλλά και κυρίω και στις δυνάμεις ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις που χωρίς καμία αμφιβολία ήταν ε, υπεύθυνοι, ε, υπέτη ή κάποιος είναι του για την ε, εξαφάνιση του επιζώντος αυτού της δικτατορίας. Επίσης θα ήταν σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, ρίξει μια ματιά στην περίπλοκη κατάσταση που ε, γνωρίζουν οι επιζώντες των ε, στρατοπέδων αυτών συγκέντρωσης, εξαφάνισης και βασανιστήριων που δυστυχώς υπήρχαν στην Αργεντινή εκείνη την εποχή. Είναι σημαντικό. Εάν η Αργεντινή, το κράτος, οι δικαστές και εκείνοι που καλούνται να διερευνήσουν αυτή την εποχή και να προστατεύουν τους επιζώντες μάρτυρες θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη το άμεσο ενδιαφέρον που δείχνει η διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το καιρό γίνονται πολλές δίκες στη χώρα μας. Και αυτό είναι κάτι που μας κάνει πολύ υπερήφανους. Ήδη πριν από έξι χρόνια ξεκίνησε αυτή η δικασία και νομίζουμε ότι θα διαρκέσει μερικά χρόνια ακόμα. Και αυτό έγινε με τη διεθνή αλληλεγγύη, με την πολιτική δράση, με τη ε, νομική και δικαστική δράση που αναπτύσσεται σε διάφορα κράτη της Ένωσης, όπως είναι η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, όπου έγιναν δίκες κατά Αργεντινών στρατιωτικών. Ενώ στην Αρχεντινή ήταν αδύνατο κάτι τέτοιο. Ήταν αδύνατο να δικαστούν οι πέτοι ακριβώς λόγω του νομικού πλαισίου ατιμορρησίας που επικρατούσε μέχρι το 2003. Και πρέπει να σας πω ότι εάν σήμερα αποδίδουμε δικαιοσύνη στην Αργεντινή και αν σήμερα είναι παράδειγμα για πολλούς οι Αργεντινοί και μπορούμε να το δανειστούμε και για τη Βερμανία και για πολλά άλλα παραδείγματα, αλλά και για τους αδελφούς μας Λατινικής Αμερικής. Ε, σκέφτομαι εδώ τη Χιλή, την Ουρουγουάη, τη Βραζιλία, το Περού, όπου έχουν την πρόθεση να δικάσουν εκείνους που μαζικά παραβίασαν τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες αυτές. Αλλά δυστυχώς ακόμα συνεχίζουν να απολαμβάνουν ατιμορρησία. Γίνονται λοιπόν πρόοδοι σε αυτή τη διαδικασία της δικαιοσύνης στην Αργεντίνα είναι, συγγνώμη, και δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι αυτό θα έχει επιπτώσεις και στις αδελφές χώρες της περιοχής. Και εδώ σκέφτομαι ακριβώς τη Χιλή που σήμερα δυστυχώς κυβερνάται εν μέρη από τους πολιτικούς κληρονόμους του ε, δικτάτορα Πινοσέτ και θέλουν να επιβάλλουν το δικό τους όραμα και τη δίκη τη θεώρηση σε σχέση με τους αγνοούμενους εκείνους που έχουν υποστεί βασανιστήρια και έχουν θανατωθεί στη χώρα. Στην Αργεντινή λοιπόν η διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντική όχι μόνο από πλευρά νομική, αλλά και θεσμικής και κυρίως πολιτικής για να ε, γράψουμε ιστορία και να συζητήσουμε για την ιστορία. Σήμερα μέρα με τη μέρα στην Αργεντινή τα μέσα ενημέρωσης ενημερώνουν τον κόσμο για τις εμπειρίες των επιζώντων που καταθέτουν ως μάρτυρες στις δίκες αυτές. Κάθε μέρα εμφανίζονται ενώπιον των δικαστηρίων και αυτό έχει αντίκτυπο στον τύπο. Και ε, σε ευαίσθητους τομείς της πολιτικής, της κοινωνίας, όπως είναι τα συνδικάτα, φοιτητές, μικρά παιδιά, έφηβοι, 15, 16, 17 ετών, συζητούν το πρόσφατο παρελθόν της Αργεντινής. Και αυτό μας γεμίζει περηφάνεια πραγματικά, γιατί για πρώτη φορά στην Αργεντινή, για πρώτη φορά τα παιδιά μας και η κοινωνία ολόκληρη ε, μαθαίνουν και γνωρίζουν ποιο ήταν το δράμα ε, των στρατοπέδων και της εξαφάνισης και των βασανιστήριων στην Αργεντινή. Και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να επιμείνουμε οι δίκες εκείνες που ξεκίνησαν σε διάφορες χώρες στην Ευρώπη να μπορέσουν να βρουν συνέχεια και να συνεχίσουν να δίνουν καρπούς. Τώρα περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ε, Αργεντινή. Δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν έχουν λήξει οι δίκες αυτές που έγιναν στην Ευρώπη κατά των Αργεντινών στρατιωτικών. Και η καρπή αυτή είναι κάτι που χρειάζονται ε, την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενημερωθεί και να ενημερώνεται σημαντικά και καθημερινά για το τι συμβαίνει στην Αργεντινή. Γιατί μπορεί να έχει δρομολογηθεί η διαδικασία, να έχει ξεκινήσει και να προχωρούμε. Είναι γεγονό, όπω είπε και ο δικαστή Ραφέκα, ότι υπάρχουν ακόμη κάποιοι θύλακε που εξακολουθούν να παραμένουν σε ατιμορρησία, όχι μόνο στην Αργεντινή, αλλά και σε άλλου τομεί και σε άλλε χώρε. Σιγά σιγά αυτά θα ανοίγουν, ε, αλλά θα υπάρξουν και αντιστάσεις και κάπου στην κοινωνία θα φανεί αυτό. Λοιπόν, γίνονται δίκες, προχωρούμε, αλλά οι κίνδυνοι δεν έχουν εξαφανιστεί. Υπάρχουν ακόμα. Η συζήτηση θα πρέπει να συνεχίσει να γίνεται. Ο αγώνας θα πρέπει να συνεχιστεί και στη χώρα μας και στην περιοχή γενικότερα. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ να εκπροσωπήσουμε με τη δική μας φωνή ε, πολλές χιλιάδες ε, θυμάτων των οικογενειών τους και όπως είπε και ο δικαστής ε, Ραφέκας και την Αργεντινή την ίδια, το κράτος. Για να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς να παρέμβει, να ακουστεί η φωνή της δημόσια για την κατάσταση αυτή. Και η κατάσταση των μαρτύρων, να δούμε τι έγινε με τον Χούλιο Λόπες, να μην ξαναεπαναληφθεί μια τέτοια περίπτωση και να καταστεί σαφές ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ η διεθνής κοινότητα να προχωρήσουν οι δίκες να ολοκληρωθούν με τρόπο σοβαρό και οι ποινές που θα επιβληθούν να ε, είναι πραγματικές ποινές και όχι εικονικές, να εκτίσουν τις ποινές τους οι ε, πέτοι. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που μας δίνετε το λόγο. Θα παραμείνουμε σε επαφή ε, για να σας ενημερώνουμε για ό,τι χρειαστεί και στο μέλλον. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Γιάνσον. Είμαι σίγουρη ότι θα ακουστούν ερωτήσεις. Θα δώσω το λόγο για ερωτήσεις. Ο πρόεδρος της ε, αντιπροσωπείας ε, για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Αργεντινής, προσπαθώ να τον τίτλο της αντιπροσωπείας αυτής, είναι η αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες με Κοσούρο. Ο, κύριο, ο πρόεδρος λοιπόν είναι εδώ για να συμμετάσχει στις ε, συζητήσεις. Πρόεδρε, λοιπόν, όποτε θέλετε να πάρετε το λόγο, είναι στη διάθεσή σα, και ούτω ή άλλω εσεί θα κλείσετε την ακρόαση αυτή. Η αλλω ε, την Πορτογαλία. Ο Λουίς πρώτα. Ίσως, ίσως θα κλεισετε την ακροαση αυτη η αννα γκομες που που προερχεται απο την πορτογαλια ο λουις θα ξεκινησει ο προεδρος της αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Μονάχα σε ένα τυπικό επίπεδο βάση της μέσης διάταξης όπως την έχω στα χέρια μου και φαντάζομαι και όλοι οι βουλευτές της ε, Επιτροπής μας. Οι παρεμβάσεις πριν από την συζήτηση και την άντληση των συμπερασμάτων Νομίζω ότι υπάρχει ακόμα κάποιο ακόμα ο οποίο θα λάβει το λόγο, ο προσβευτή τη Αργεντινή, ο κ. Βλέτνικοφ, ο οποίο είναι παρόν. Προτού καταλήξω εγώ σε συμπεράσματα, νομίζω θα ήταν πιο πρόσφορο να καταλήξει η συζήτηση με την παρέμβαση και του πρεσβευτή της Αργεντινής και μόνο μετά εγώ να λάβω το λόγο για τα συμπεράσματα. Ε, θα, σας... θα δεχθούμε τη συμβουλή σα, Ούτως ή άλλως σκόπευα να δώσω το λόγο και στον πρέσβη. Κύριε Πρεσβευτά, μπορείτε να πάρετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για το γεγονός ότι ο Υφυπουργό Εξωτερικών επισκέφτηκε στο γραφείο μου πριν από λίγε μέρε και μου έδωσε την ευκαιρία να καταλάβω πόσο πολύ έχει εμπλακεί η χώρα σα σε αυτή τη διαδικασία προ τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα συμπληρώσω λίγο τις ε, πληροφορίε. την ενημέρωση των δύο συμπατριωτών. Ο δικαστής Ραφέκας και ο κύριος Γιάνσον θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ στη θέση της Αργεντινής σε αυτά τα θέματα ε, σε ένα διεθνές πλαίσιο. Όπως σίγουρα γνωρίζετε πολλοί από εσά, η Αργεντινή και η Ευρώπη έχουν μακρά παράδοση φιλίας και ε, αμοιβαίων σχέσεων μοιραζόμαστε ιδέες, πολιτισμό, επενδύσεις, εμπόριο, καθώς και εκατομμύρια εκατομμυρίων Ευρωπαίοι ε, ήρθαν στη χώρα μου και τις δέχτηκε η Αργεντινή από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ου. και το αντίστροφο ε, κατέφυγαν στην Ευρώπη και τους δέχτηκε η Αργεντινή μετά τη δικτατορία και λόγω οικονομικών προβλημάτων. Έχουμε λοιπόν μια συναντήληψη θα έλεγα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ζητήματα όπως είναι η προστασία της δημοκρατίας, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση της ξενοφοβίας καθώς επίσης και των διακρίσεων, η ε, κατάργηση της ατιμορρησίας και συμμετοχή στα πράγματα της κοινωνίας των πολιτών. Σε όλα αυτά τα θέματα η Αργεντινή θεωρεί ότι είναι απόλυτα οικουμενικά θεμελιώδη δικαιώματα. Εμείς από την Αργεντινή σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να διαφέρουμε σε θέματα οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά γιατί ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης κάθε χώρα γνωρίζει τη στρατηγική καταρτίζει. Αλλά σε αυτά τα θέματα που μας απασχολούν τώρα θεωρούμε ότι τα δικαιώματα είναι απόλυτα αδιαπραγμάτευτα και δεν θα πρέπει να υπάρχουν διαφορές στην ερμηνεία. Για την Αργεντινή, η καταπολέμηση της ατιμορρησίας και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ε, κεντρική ιδέα της κοινωνίας μας και βασική πυλώνες της σημερινής κυβέρνησης. Η αλήθεια, η μνήμη, η δικαιοσύνη, η αποκατάσταση είναι βάσεις για να οικοδομηθεί η πλήρης δημοκρατία και ε, γερή δημοκρατία. Αυτή τη θέση την ενέκριναν, την υιοθέτησαν και οι τρεις εξουσίες στη δημοκρατία μας, που είναι η νομοθετική εξουσία, η δικαστική εξουσία και η εκτελεστική εξουσία. Οι δίκες για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας είναι πολιτική του κράτους, όπως πρόσφατα ενέκρινε η Βουλή μας. Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η πιο πρόσφατη δικτατορία μας σημάδεψε. Και εσείς οι Ευρωπαίοι γνωρίσατε πολλές ε, χούντες και καταφέρατε από αυτή την τρομερή σας εμπειρία να οικοδομήσετε μια δημοκρατία. Και εμείς οι ίδιοι οικοδομούμε τη δημοκρατία μας από το 1983 και μετά. Αργεντίνα, η... η Αργεντινή και η Ευρωπαϊκή Ένωση από το Δεκέμβριο του 2008 έχουν ε, εγκαθιδρύσει ένα πολιτικό διάλογο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουν ήδη πολλές συναντήσεις με στόχο το συντονισμό της κοινή δράσης στα διεθνή φόρα, ιδιαίτερα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και τη Γενική Συνέλευση στη Νέα Υόρκη. Προφανώς και στις διμερείς μας σχέσεις επίσης. Ιδιαίτερος συμφωνούμε για την πρόθεση της κύρωσης της σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από την καταναγκαστική εξαφάνιση. Στην Αργεντινή και στη Γαλλία, αλλά χρειάζεται ακόμα για να τεθεί σε ισχύ και άλλη μία κύρωση. Επίσης, έχουμε κοινή δράση ε, Αργεντινή και Ευρώπη για την ε, ε, εξάλληψη της θανατικής ποινής και την καταπολέμηση τη ατιμορρυσία στα πιο σοβαρά εγκλήματα στο διεθνέ δίκαιο και υποστηρίζουμε εδώ το έργο του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου. Αυτά είναι λίγα μόνο παραδείγματα της τόσο γόνιμης συνεργασίας που έχουμε γιατί μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα σε αυτά τα θέματα που είναι τόσο θεμελιώδη και τόσο κομβικά για την ενίσχυση του δημοκρατικού συστήματος. Επιπλέον, η Αργεντινή προωθεί πρωτοβουλίες για το δικαίωμα στην αλήθεια και ε, να χρησιμοποιούμε το γενετικό υλικό στην ιατροδικαστική για να ε, διαπιστώνουμε, εξακριβώνουμε ακριβώς τα στοιχεία και ποια πρόσωπα υπέστησαν αυτά τα βαρύτατα εγκλήματα. Και στις δύο περιπτώσεις η χώρα μας υπέβαλε ψηφίσματα που εγκρίθηκαν ομόφωνα ε, στην Επιτροπή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με μια σειρά άλλες χώρες που μας υποστήριξαν. Επίσης, μια που εδώ είμαστε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρέπει να πω ότι η Αργεντινή Επιπροεδρία στις, στην Λατινική Αμερική και Καραϊβική, στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι την πρόσφατη σύνοδο που έγινε στη Μαδρίτη τον περασμένο Μάιο, η Αργεντινή ανέκαθεν πίεζε και επιθυμούσε για να έχει ένα διάλογο γόνιμο και σε βάθος με όλη τη ε, Λατινική Αμερική και την Καραϊβική και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι πέρυσι επιτύχαμε οι δύο περιφέρειες, τα δύο μέρη να ξεκινήσουν ένα διάλογο που θα συνεδριάζει κάθε δύο-τρεις μήνες και εκεί θα συζητούμε και θα λύνουμε τα προβλήματα που έχουν οι μετανάστες από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική στην Ευρώπη. Για να έχετε μια ιδέα, έτσι, μια τάξη μεγέθου είναι 6 με 8 εκατομμύρια ε, μετανάστες αυτοί. Τολμώ να πω ότι η Αργεντινή σε αυτό το θέμα της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ε, πραγματικά παράδειγμα, υπόδειγμα για την περιοχή σε αυτά τα θέματα και κυρίως στην καταπολέμηση της ατιμορρησίας. Στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλους πολυμερείς οργανισμούς ε, είμαστε σε θέση να συνεργαζόμαστε ε, μεταξύ μας και ε, υποστηρίζοντας το Διεθνές Πενικό Δικαστήριο. Συμπερασματικά λέγω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε στα θετικά στους κοινού αγώνες για τη δημοκρατία, για το κράτος δικαίου, για την πρόθεση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την κατάργηση της ανατικής ποινή για την αποδοχή της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε θέματα διεθνούς δικαίου και για την ε, αστυνομική συνεργασία σε αυτά τα θέματα. Επίσης μπορούμε να συνεργαζόμαστε ε, κατά της ατιμωρησίας, κατά των διακρίσεων, κατά της ξενοφοβίας, κατά κάθε είδους ε, αδιαλαξίας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Thank you very much for your contribution. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη και τώρα θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους για να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Η κυρία Γκόμες, βεβαίως πρώτη και καλύτερη. Είναι πορτοκαλίδα και κάτι ξέρει από δικτατορίες. Como Σαν δείγμα της εκτίμησής μου για τους καλεσμένους μας από την Αργεντίνα, την Αργεντινή και, τους, και τον προσβευτή της Ισπανίας, θα μιλήσω σε σπανικά. Πιστεύω ότι πράγματι η Αργεντινή είναι ένα καταπληκτικό παράδειγμα για την ανθρωπότητα και για εμάς τους ίδιους, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχομαι από μία από αυτές τις χώρες που πέρασε μια δικτατορία, που πέρασε μια μεγάλη μακρά χρονική δικτατορία, την Πορτογαλία. Θα ήθελα η χώρα μου να είχε περάσει τη φάση αυτή της δικαιοσύνης που βλέπουμε σήμερα στην Αργεντινή. Πολλά από τα προβλήματα που έχουμε σήμερα δεν θα είχαν προκύψει αν η δικαιοσύνη είχε κάνει το έργο της όπως πράγματι λαμβάνει η χώρα σήμερα στην Αργεντινή. Εγώ παρακολούσα από πολύ κοντά όλη αυτή τη διαδικασία μέσα από τις δομές του ΟΗΕ στην προηγούμενη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και για μένα πρέπει να πω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό το έργο αυτό της Αργεντινής από τη στιγμή που ξεφορτώθηκε τη δικτατορία η προσπάθεια απόδοσης δικαιοσύνης και ανακάλυψης της αλήθειας στη χώρα αυτή, αλλά όλα αυτά προς όφελος της οικουμενικής δικαιοσύνης, όχι μόνο με τη δημιουργία μηχανισμούς όπως η ομάδα εργασίας για τους αγνοούμενους, για τα άτομα που εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, Όλες αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν που δημιουργήθηκε από τη δικτατορία την αρχή της Αργεντινής αυτός ο καταχθόνιος μηχανισμός εξαφάνισης ατόμων που φοβάμαι ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τέτοιοι μηχανισμοί υπάρχουν και σε πολλές χώρες ακόμα, άλλες χώρες ακόμα και σήμερα αλλά κυρίως μας ενδιέφερε η δέσμευση της Αργεντινής σε διάφορα διεθνή φόρα και σε πολλές καταστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο όπου λαμβάνουν χώρα παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι κάτι το οποίο είναι κοινό σε όλες τις χώρες που έχουν βγει από δικατορίες και έχουν προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Αργεντινή πάντα υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει απόδοση δικαιοσύνη. Στην περίπτωση Βιρμανίας που συζητούσαμε σήμερα το πρωί, θυμάμαι αυτά τα οποία ελέγχθησαν σήμερα το πρωί, ότι στη δεκαετία του 80 υπήρξαν αντίστοιχε περιπτώσει σε πολλές χώρες του κόσμου και επομένω είναι απαραίτητο να υπάρξει υποστήριξη για τις πρωτοβουλίες των Ευρωπαίων σε σχέση με τη, με τη Βερμανία. Η Αργεντινή λοιπόν ήταν η πρώτη, ο πρώτος σύμμαχός μας σε αυτή την προσπάθεια καταπολέμησης της ατιμορρησίας. Να υπάρξει δικαιοσύνη λοιπόν σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλω να τονίσω ότι για τη χώρα μου υπήρξε πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίες έχουν συμβεί στη χώρα μας. Έχουμε μια ακόμα, ένα ακόμα παράδειγμα, την περίπτωση του Ανατολικού Τιμόρ που μπορέσαμε στην περίπτωση αυτή να έχουμε την υποστήριξη της Αργεντινής. Νομίζω λοιπόν ότι η κατάσταση της Αργεντινής και όλες οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται για την αποκατάσταση του δικαίου είναι πολύ σημαντικές και ένα σημαντικό παράδειγμα και για άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Οι εκπρόσωποι της Αργεντινής νομίζω ότι δεν ανέφεραν μια περίπτωση που εμένα με ενδιέφερε πάρα πολύ και όπου πιστεύω ότι μπορούμε να, να πάρουμε διδάγματα από την κατάσταση της Αργεντινής είναι η τρέχουσα κατάσταση στην Κολομβία όπου υπάρχουν γενναίοι δικαστικοί οι οποίοι όμως δεν έχουν την απαραίτητη πολιτική και θεσμική υποστήριξη. Κάτι το οποίο όμως βλέπουμε να υπάρχει σήμερα στην Αργεντινή. Ευχαριστώ. Κάτι ακόμα το οποίο ήθελα να πω. Δεν ήθελα να ξεχάσω ότι η Αργεντινή είναι και ένα παράδειγμα όταν στην περίπτωση μιας άλλης χώρας που πολιτιστικά και γεωγραφικά ε, είναι κοντά σε μια χώρα πολιτιστικά μάλλον είναι κοντά στην ε, Αργεντινή, στην Ισπανία, μια χώρα που είναι γεωγραφικά κοντά στη δική μας, στην Πορτογαλία. Υπάρχει μια αντιμετώπιση που εμποδίζει να ανακαλυφθούν οι αγνοούμενοι και οι νεκροί του εμφύλιου πολέμου στην Ισπανία και όπου υπάρχει μια τόσο αρνητική στάση απέναντι στη γενναία προσπάθεια του Μπαλτασάρ Καρσόν. Ευχαριστώ. Η κυρία Κίλ Νίλσαν ε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές. Νομίζω, εγώ τουλάχιστον βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την παρουσίασή τους. Ε, θέλω να θέσω κάποιες ερωτήσεις. Κάποια θέματα βέβαια τα έχετε ήδη θίξει. Το βασικό ερώτημα είναι αυτό που συμβαίνει στην Αργεντινή, τι επίπτωση έχει στις άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, αλλά και πιο πέρα, στις πιο μακρινές χώρες. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, πώς θα μπορέσουμε να γενικεύσουμε αυτή την πρακτική, η οποία είναι πραγματικά παραδειγματική. Τι περιμένετε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από εμά. Ερχόμενοι εδώ, σκεφτόμουν αυτό το ερώτημα. Ε, είναι σημαντικό να σταθούμε λίγο σε αυτό το σημείο σήμερα. Και τέλος, ε, μια άλλη ερώτηση. Μιλάτε για αυτές τις δίκες που λαμβάνουν χώρα. Υπάρχει πιθανότητα πραγματικά να καταδικαστούν οι ένοχοι και τι είδου ε, καταδίκες περιμένετε ότι θα, θα υπάρξουν. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ. Η κυρία Σινκλέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας, ευχαριστώ τον πρεσβευτή που παρουσίασαν τόσο συνολικά το θέμα που είναι δύσκολο να ε, βρω ερωτήσεις. Πέρυσι επισκέφθηκα την Αργεντινή, είναι μια θαυμάσια υπέροχη χώρα, πολύ ζωντανή και νομίζω ότι είναι στραμμένη προς το μέλλον, σε ένα πιο θετικό μέλλον. Ε, σκόπευα να ξαναπάω ε, τον επόμενο μήνα, αλλά χρειάστηκε να την αναβάλω αυτή την ε, επίσκεψη. Πάντως η αλλαγή ε, εξαπλώνεται σε όλη τη Λατινική Αμερική, με μπροστά, μπροστάρι όμως την Αργεντινή με αυτές τις δίκες. Αυτό αποδίδει δικαιοσύνη στα θύματα. Είναι παράδειγμα και για τη Βυρμανία, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα κρυφτούν, θα δικαστούν τελικά σε 10-15 χρόνια έστω. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, είναι... Σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε προς αυτήν την κατεύθυνση. Εγώ ξέρετε ότι δεν υποστηρίζω πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε, με κάθε ευκαιρία την επικρίνω. Αλλά κάτι θετικό είναι ε, το βραβείο Ζαχάροφ. Ε, μη, νικητές του βραβείου αυτού οι μητέρες της πλατείας του Μαΐου. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνουμε και εμείς τη διαδικασία ε, που υπάρχει στην Αργεντινή. Έχω πολλούς φίλους στην Αργεντινή, είμαι σε επαφή μαζί τους, μέσα του facebook κτλ. Και ένα πράγμα που διαισθάνομαι είναι ότι δεν τους αρέσουν τα διδάγματα από τις πρώην απεικιοκρατικές ε, δυνάμεις. Διερωτώ με, λοιπόν, ότι ναι μεν θέλουμε να σας υποστηρίξουμε, αλλά δεν θέλω σε καμία περίπτωση να πιστέψετε ότι εμείς ε, κάνουμε κηρύγματα, από καθέδρας ειδικά. Όχι, θέλω να μιλήσουμε επίσης όρις. Ευχαριστώ κυρία Σινκλέρ. Τώρα, ο πρόεδρος αντιπροσωπείας ε, με τις χώρες του Μερκοσούρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την πρωτοβουλία που ανέλαβε να θέσει αυτό το θέμα στη μέση διάταξη για την καταπολέμηση της ατιμορρησίας και το παράδειγμα της Αργεντινής. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και κυρίως το δικαστή ε, Ραφέκας, ε, το κύριο Γιανσόν και τον πρέσβη ε, για την ενημέρωση που μας έκαναν. Αυτό τι σημαίνει. Ότι μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα από τα στοιχεία αυτά που μαθαίνουμε από τη συζήτηση. Και οι τρεις συνάδελφοι ευρωβουλευτές που μίλησαν πριν από μένα ήρθαν να συμπληρώσουν αυτά που λέει. Κατά την άποψή μου, με την υποστήριξη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και διατρανώνοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε την ατιμορρησία για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και με τη συμπερίληψη κοινή νόμης να διαπαιδαγωγήσουμε έτσι την κοινή γνώμη και θα αναφερθώ στη συνέχεια σε αυτό, να υποστηρίξει όλους τους ενδιαφερομένους σε αυτή την ε, ε, υπόθεση, αυτόν τον αγώνα, Κυβερνητικέ και μη οργανώσεις ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κόμματα, μέσα ενημέρωση, συνδικάτα που μέσα από τόσες δυσκολίες κατάφεραν να δημιουργήσουν κάτι που πιάνει τόπο και Μαθαίνει ο λαός από αυτό. Η Αργεντινή μας δίνει το παράδειγμα για το πώς θα πρέπει να προχωρούμε. Και είναι και προηγούμενο. Μακάρι όλες οι χώρες που υπέστησαν ή που υφίστανται σήμερα στον κόσμο δικτατορίες και καταπιεστικά, κατασταλτικά καθεστώτα που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, μακάρι λέγω να έχουν την ίδια αντιμετώπιση στη συνέχεια δίωξη στη δικαιοσύνη, επαγρύπνηση και καταδίκη των υπετίων. Ο 20ος αιώνας στην Ευρώπη, το είπε η κυρία Σενκλέρ έμεσα, τουλάχιστον τα πρώτα 50 χρόνια δεν ήταν ε, υποδειγματικά ακριβώς. Κυριαρχούσαν οι απολυταρχισμοί, οι φασίστες, οι σταλινικοί. Και είχαμε χούντες, δικτατορίες, καταπιεστικά καθεστώτα με δεκάδες χιλιάδες και εκατομμύρια νεκρούς στο ολοκαύτωμα, με ε, διώξεις, ε, δολοφονίες, βασανιστήρια. Αλλά στο δεύτερο μέρος του 20ου αιώνα παρέμειναν κάποιες δικτατορίες, όπως είπε η κυρία Γκόμες, στην ίδια μου τη χώρα, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, αργότερα οι συνταγματάρχες στην Ελλάδα, η Χούντα των Συνταγματαρχών. Συμφωνώ με την κυρία Γκόμες απολύτως. Ούτε στην Ισπανία δεν καταπολεμήθηκε η ατιμορρησία έτσι με συνέπεια και μέχρι τέλους. Γιατί προηγουμένως γι' αυτό σας μίλησα για τη διαπαιδαγώγηση του πληθυσμού. διαφοέρει η αντίληψη, η αίσθηση του λαού από εποχή σε εποχή. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 όταν έπεσε η Χούντα στην Ισπανία και πέρασαμε στη Δημοκρατία δεν ε, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την τιμωρία εκείνων που ήταν υπεύθυνοι και μετά από τον εμφύλιο πόλεμο. Και μιλώ για την οπισθοφυλακή προσοχή, όχι εκείνους που έχασαν τη ζωή στο μέτωπο. Και μέχρι την αρχή της δεκαετίας του 50 υφίστανται διωγμούς και βασανισμούς και αργότερα από πλευράς ποινική και δικαστικής ήταν ακόμα πιο δύσκολο γιατί είχαν περάσει τα χρόνια πια. Και εγώ βέβαια δομικός δεν είμαι, αλλά το ποινικό δίκαιο απαιτεί να ζει να είναι εν ζωή ο ε, υπέτειος. Αυτή τη στιγμή εκλείψει ο ενδιαφερόμενο, έχει πεθάνει, δεν δικάζεται στο ποινικό δίκαιο. Τον δικάζει η ιστορία βεβαίω, αλλά δεν τον δικάζει το ποινικό δίκαιο. Ε, και ο ε, δικαστής Γκαρθών, που ήταν τότε ε, δικαστής στην Αουδιένθια Νασιονάλ, ε, γιατί 140.000 ε, θύματα και αγνοούμενοι του εμφυλίου πολέμου ε, βρίσκονται θαμένοι σε καινοτάφια, σε άγνωστα σημεία και δεν έχουν βρεθεί. Και ε, τι κάνει η κυβέρνηση στη συνέχεια, ε, ε τον διώκει, τον δικαστή Γκαρσόν για κατάχρηση εξουσίας. Πράγμα που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος στην Ισπανία, που υποστηρίζει τα θύματα του φραγκισμού. Ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να φέρουμε σε αίσιο πέρα σε αυτή την υπόθεση. Και μια τελευταία παρατήρηση. Επιμένω πάρα πολύ ότι είναι πολύ σημαντική η αίσθηση της κοινή γνώμης. Δεν είναι ίδιες οι εποχές. Το 1983 ο πρόεδρος Αλφονσίν στην Αργεντινή ε, κάθισε στο εδόλιο τρεις στρατιωτικές ε, χούντες ε, υπετίους πραξικομάτων. Δεν έγινε αυτό πουθενά μέχρι τότε. Από εκεί και πέρα ε, έγιναν κάποιες προσπάθειες να ε, κλείσει οριστικά αυτό το θέμα ο φάκελος της δικτατορίας αλλά τα τελευταία χρόνια ε, ξανά άνοιξε αυτό το θέμα για να ξεπεραστεί η Αλλά Πρέπει να το πω αυτό. Ο πρόεδρος Αλφωσίν μετά το τέλος της δικτατορίας ε, υποστήριξε πάρα πολύ και υπηρέτησε πάρα πολύ αυτή την ιδέα και αυτή τη φιλοσοφία. Τέλος, Πρόεδρε, πρέπει να πούμε ότι είναι οικουμενική η δικαιοσύνη, είναι παγκόσμια, γιατί υπάρχουν πολλοί εχθροί της που θέλουν να την καταργήσουν και είναι βασικό στοιχείο για την καταπολέμηση της ατιμορρησίας που επαναλαμβάνω είναι υπόδειγμα η Αργεντινή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Γιάννης για τα πολύ κέρια σχόλιά σας. Είμαι σίγουρη ότι θα ακούσουμε τις απαντήσεις από των τριών προσκεκλημένων μας. Και ίσως και κάποιες άλλες παρατηρήσεις. Τώρα, να σας πω κάτι, ότι συχνά εδώ στην Υποεπιτροπή μας πλησιάζουν τα θύματα διωγμών, φρικαλαιοτήτων κτλ. Και φυσικά είμαστε ένα πολιτικό όργανο, δεν είμαστε δικαστικό όργανο. Αλλά αυτό που με απασχολεί είναι το εξή. Τι μπορούμε εμεί να προσφέρουμε σε αυτά τα θύματα ε, του Βορείου Καυκάσου, της Τριλάνκας και άλλων ε, σημείων του πλανήτη, Βόρειας Κορέας, Βυρμανίας, θύματα φρικαλαιοτήτων, όπου σε ορισμένε χώρε τουλάχιστον τα θύματα συλλέγουν ε, ντοκουμέντα, τεκμήρια για σοβαρότατες παραβιάσεις ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τα εγκλήματα αυτά, του δικαιώματο στη ζωή κτλ. Έχετε κάποιες ιδέες, ε, η Αργεντινή μπορεί να μας βοηθήσει, πώς εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τις ομάδες αυτές θυμάτων που θέλουν να κρατήσουν αυτά τα ντοκουμέντα ε, που αποδεικνύουν την ενοχή των δολοφόνων, των διοκτών κτλ. Μέχρι την εποχή που θα διωχθούν και θα εμφανιστούν ενώπιον δικαστηρίου. Θα σας ήμουν ευγνώμων για τις απαντήσεις, γιατί συχνά έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους που βρίσκονται σε τέτοια επαχθή κατάσταση και συχνά απειλείται η ζωή τους. Γιατί φυσικά κάποιες ε, δυνάμεις ασφαλείας ή κάποιες κυβερνήσεις κάνουν ό,τι μπορούν για να τους φημώσουν και να μην δουν το φως τέτοια ντοκουμέντα. Και φυσικά διώκουν τους ανθρώπους οι οποίοι επιδίδονται σε τέτοιες δραστηριότητες. Ας ακούσουμε λοιπόν ακόμα μια φορά ε, καταρχήν το δικαστή Ραφέκας. Ε, τι έχει να μας πει για αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να σας απαντήσω σύντομα, κυρία Πρόεδρε. Για αυτή την ανησυχία που εκφράζεται. Θέλω να επαναλάβω καταρχήν ότι είναι πολύ σημαντικό για αυτή τη διαδικασία που είναι εξελίξει στην Αργεντινή, για την δικαιοσύνη, ε, για τις δίκες, αλλά κυρίως για τα θύματα της Αργεντινής, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν μια δημόσια δήλωση υποστήριξης αυτής της διαδικασίας. Αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις και άμεσα στην Αργεντινή αλλά και έμεσα στις υπόλοιπες χώρες της περιοχής της Λατινικής Αμερικής δηλαδή, όπου υπάρχουν ε, κάποιες αμφιταλαντεύσεις των κυβερνήσεων για το αν θα πρέπει να κάνουν αυτό το πίδημα προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως το έκανε η Αργεντινή τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναφέρουν την Αργεντινή και να γνωρίζουν τα τεκτενόμενα, να γνωρίζουν ε, τι γίνεται σε νομοθετικό επίπεδο, σε δικαστικό επίπεδο, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο, να ενδιαφερθούν για τα τεκτενόμενα. Οι ε, ευρωβουλευτές, μόνο και μόνο με την επίσκεψή τους στην χώρα μας, θα έχουν τεράστια ε, επιρροή μέσω της δημοσιότητας που θα δοθεί. Επίσης θα πρέπει να υπάρξουν από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης προγράμματα οικονομικής βοήθειας ή ενίσχυσης των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Γνωρίζουμε την τεράστια εμπειρία που έχει η Ευρώπη σε τέτοιου είδους πρακτικές, σε τέτοιου είδους διασκέψεις, συνέδρια κτλ. Και μπορείτε να μας βοηθήσετε λοιπόν προς αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα να απαντήσω στις υπόλοιπες ερωτήσεις ε, των υπολείπων ομιλητών. Τι να απαντήσω στο ερώτημα αν η πολιτική αυτή της Αργεντινής για την δικαιοσύνη και την ε, μνήμη έχει επηρεάσει την υπόλοιπη περιοχή. Η προσωπική μου γνώμη είναι δεν προκάλεσε την, την αναστάτωση. Δεν επηρέασε τα πράγματα όπως θα έπρεπε να τα επηρεάσει. Εμείς ήμασταν αισιόδοξοι και πιστεύαμε ότι θα υπάρξει μια έτσι, μεταδοτικότητα ας πούμε, στις ε, αδερφές χώρες, ιδίως στην Ουρουγουάη, στη Χιλή, στην Παραγουάη. Θα μεταδοθεί αυτή η διαδικασία, θα μεταλαμπαδευτεί. Αλλά αυτή η μεταλαμπάδευση δεν έχει σημειωθεί. Δεν έγινε τίποτα το απτό. Πρέπει βεβαίως να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να το επιτύχουμε. Η Αργεντινή και δημόσια αλλά και μέσω των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, εργάζεται ούτως ώστε οι χώρες αυτές να ανοίξουν τα μάτια, να κινηθούν προς αυτή τη διαδικασία δικαιοσύνης ε, και μνήμης και δικαιοσύνης. Αλλά αμφιταλαντεύονται οι χώρες αυτές. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουν αυτό το βήμα. Νομίζω ότι και προ αυτή την κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει. Φερρυπίν, να οργανώνει συνεδριάσει, εργασίες ε, επίσημες για αυτά τα θέματα και να καλεί και τις διάφορες χώρες. Και να έρχονται Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες και Αργεντινοί ή, εν πάση περιπτώσει, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διοργανώνται τέτοια σεμινάρια, ε, συνέδρια, γιατί θα είχαν τεράστια σημασία, έστω και συμβολική. Και τέλος, για να απαντήσω στην κυρία Γκόμες, για τι είδους ε, καταδίκες περιμένουμε, είναι ανάλογες οι καταδίκες αυτές με τα εγκλήματα που διεπράχθησαν. Και σε κάθε περίπτωση βλέπουμε τα εγκλήματα του κάθε κατηγορούμενου. Μερικές φορές έχουμε σοβαρότατα εγκλήματα, ανθρωποκτονίες, ε, βασανιστήρια. Σε αυτή την περίπτωση η ποινή θα είναι η μέγιστη που προβλέπει ο νόμος. Ε, είναι δηλαδή σόβια δεσμά. Σε άλλες περιοχές, περιπτώσεις θα είναι μία ποινή φυλάκισης ε, που φτάνει μέχρι και 25 χρόνια. Σε άλλες περιπτώσεις δε, αν υπάρχει συνενοχή ή αν έχουν διαπραχθεί αδικήματα, απλώς και όχι εγκλήματα, οι ποινές είναι μικρότερες. Επαναλαμβάνω όμως, στις δίκες αυτές που λαμβάνουν χώρα στην Αργεντινή τα δικαστήρια αυτά είναι αστικά δικαστήρια, τα οποία εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία και το γράμμα του νόμου. Εμείς δεν επηρεάζουμε τα αστικά δικαστήρια. Άλλη ποινική διαδικασία, άλλη αστική. Έχουμε εξαλείψει την θανατική ποινή στην Αργεντινή. Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι κατηγορούμενοι απολάβουν όλων των δικαιωμάτων τους ανάλογα με το είδος των αδικημάτων που έχουν διαπράξει. Μετά έχουν τα δικαιώματα δηλαδή που προβλέπονται από τον νόμο για τους φυλακισμένους ή τους υπόδικους. Ευχαριστώ κύριος Γιανσόν. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τα όσα είπε μόλις ο δικαστής Ραφέκας. Θέλω μόνο να προσθέσω κάτι για τον αντίκτυπο που έχει σε άλλες χώρες και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο στοιχεία μόνο. Αφενός. Εδώ σκέφτομαι κυρίως τους δικαστές, τους εισαγγελείς. Θέλω να κάνω μια παρένθεση και να τονίσω ότι δυστυχώς σήμερα ένα τμήμα της δικαστικής εξουσίας, ένα μέρος των δικαστών στη χώρα, εξακολουθούν να βλέπουν με άλλη ματιά ε, τα πράγματα. Είναι ευνοϊκή προς την ατιμορρησία. Σήμερα βέβαια επειδή ε, δεν μπορούν, δεν εκφράζονται, αλλά όταν μπορέσουν θα εκφραστούν προς την κατεύθυνση αυτή. Τα τελευταία χρόνια όταν έλαβαν ε, γνώση και κατάλαβαν ότι θα προχωρούσαν αυτές οι δίκες, πολλοί ε, δικαστές παρετήθηκαν πάρα πολύ ε, και ζήτησαν και πρόορη συνταξιοδότηση. <laughs> Γιατί και έτσι καταλάβαμε πώς και η δικαστική εξουσία ήταν στην υπηρεσία ε, των βασανιστήριων και της εξαφάνισης. Και σήμερα υπάρχουν και δικαστές που δικάζονται και ε, έχουν στέρηση της ελευθερίας τους ακριβώς για αυτό το λόγο. Λοιπόν, σε αυτές τις ακροματικές διαδικασίες κάθε μέρα στις δίκες στη χώρα μας η παρουσία, η συμμετοχή, η άμεση επικοινωνία και διπλωματών ε, είναι ενδεικτική. Πολλές φορές συμμετείχε ο πρέσβης Γαλλικής Δημοκρατίας ή μέλη διπλωματικού σώματος εκπροσώπησης της ε, ε, ε, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τη Γερμανία και τη Ισπανία. Πολλοί πρέσβοι, πολλοί ε, διπλωμάτε έρχονται προσωπικά στα δικαστήρια, στην ακροματική διαδικασία, συζητούν με τους δικαστές, με τους εισαγγελεί. Αυτό δεν είναι ίσονο σημασία γιατί οι δικαστέ το προσέχουν αυτό, το σημειώνουν. Και εκείνοι που δεν επιθυμούν αυτέ τι δίκες θα πειθαρχήσουν, θα συμμορφωθούν. Αυτό μας χρειάζεται. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνει η ευρωπαϊκή κοινότητα και μεταξύ άλλων οργάνων ε, θεσμικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Συμμερίζομαι ε, πλήρω αυτό που είπε ο δικαστή Ραφέκα προηγουμένω. Υπάρχουν διάφορε δράσει στι οποίε μπορείτε να προβείτε για να βοηθήσετε μαζί με άλλε χώρε, αλλά και μέσω των δικών σα εκπροσώπων. Προσωπικά να κάνουν διαβήματα στην κυβέρνηση, δημόσιε δηλώσει. Γιατί ακόμα και αν αντίπαλοι είναι μικροί σε αριθμό περιορισμένοι, έχουν μεγάλη εξουσία. Και ε, ακούγεται η φωνή τους ε, σε κάποια μέσα ενημέρωση, σε κάποιες εκθέσεις. Θα πρέπει λοιπόν να απομονωθούν αυτοί οι δικαστές και κάποιοι πολιτικοί ηγέτες. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή είναι πολύ λίγοι, αλλά θα πρέπει να ε, καταλάβουμε ότι μπορεί να αυξηθούν σε λίγους μήνες. Και όπως είπε και ο βουλευτής κύριος Γενιές, αυτό εξαρτάται ε, από την κοινή γνώμη. Γι' αυτό θέλουμε να ενημερώνουμε και την κοινή γνώμη και να συνειδητοποιεί τι γίνεται με τη δικαιοσύνη. Μπορεί σήμερα να είναι παράδειγμα η Αργεντινή, ότι αφού είναι παραδειγματική εμείς τι να κάνουμε ενώ σε άλλα μέρη του κόσμου όπως στην Κολομβία και σε τόσα άλλα ε, βιάζονται και καταπατώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μα ακριβώ γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι παράδειγμα η στάση μας, πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα πρέπει να το υποστηρίξει αυτό. Γιατί αν πέσει αυτό το παράδειγμα θα γρεμιστεί το σύμπαν. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα πια ούτε στην Κολομβία, ούτε στη Χιλή, ούτε στη Βιρμανία, ούτε στην Αφρική. Ε, ε, τίποτα δεν μπορούν να κάνουν οι υπόλοιποι που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα αν καταπέσει το παράδειγμα. Για μας λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω και κάτι που λέω τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε μια ε, που επέζησε και ήρθε να καταθέσει το δικαστήριο στην Αργεντινή ως μάρτυρας σε μια ακροματική διαδικασία και ε, ενώπιον του δικαστού Ραφέκας ε, για εγκλήματα που έγιναν σε ένα παράνομο κρατητήριο ονόματι Ορλέτη. 20 μέρες τη κρατούσαν εκεί και τη βασάνισαν στο Ορλέτη. Τη γυναίκα αυτή από την Ουρουγουάη που μετά παράνομα την έστειλαν στη χώρα της όπου επίσης τη βασάνισαν μήνες ολόκληρους και έλεγε στους αργεντινούς δικαστές η κυρία αυτή Μου κάνει εντύπωση που έρχομαι εδώ και για πρώτη φορά ε, ένας δικαστής είναι πρόθυμος να ακούσει την πείρα μου και λυπάμαι που ε, είναι Αργεντινός και όχι Ουρουγουάιος. Μπορώ να μιλήσω για τις 20 μέρες αυτά που υπέστησα στην Αργεντινή, αλλά για αυτά που έζησα στην Ουρουγουάη δεν έχω πουθενά να μιλήσω. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το ακούμε από το στόμα το ίδιο μιας ε, ε επιζώσας. Ε, Χιλή λοιπόν, Παραγουάη, Ουρουάη και άλλες χώρες. Θα επαναληφθεί η εμπειρία. Είναι γεγονός αυτό που λέει ο Ραφέκα. Σε κάθε χώρα αυτό δεν ε, μετατρέπεται και σε πολιτική βούληση. Αλλά εγώ είμαι αισιόδοξη ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Αλλά θα πρέπει γι' αυτό ακριβώς το λόγο να υποστηρίξουμε το παράδειγμα της Αργεντινής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δίνω το λόγο στον πρεσβευτή τώρα τη Αργεντινή. σας ευχαριστώ πολύ ο πρεσβευτής. Απαντών και εγώ στην ερώτηση για το τι θα μπορούσε να γίνει, πώς θα μπορούσε πραγματικά να βοηθήσουμε την Αργεντινή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι καταρχήν θα πρέπει να διευρυνθεί και να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ Αργεντινής και Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μπορέσουμε έτσι να εξασφαλίσουμε στα διεθνή φόρα συγκεκριμένα στα Ενωμένα Έθνη, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να αντιμετωπιστεί το θέμα της ε, προάσπισης της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται να το αντιμετωπίσουμε σε βάθος και με μεγάλη σοβαρότητα. Για το τι μπορεί να πράξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με αυτό το θέμα για να βοηθήσει την Αργεντινή Νομίζω ότι όπως είπε και ο δικαστής ε, κ. Ραφέκας, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να εκδώσει ένα ψήφισμα το οποίο καταγράφει τις πρόοδους που έχουν επέλθει. Αυτό δεν θα ήταν αρνητικό. Αλλά υπενθυμίζω ότι η χώρα μας είναι μια κυρίαρχη χώρα όπου <clears throat> οι εξουσίες λειτουργούν ανεξάρτητα ημέν από τις δε και εμείς ως Αργεντινοί πέραν ορισμένων γκρουπούσκουλων της δεξιάς που έχουν συνεργαστεί ενεργά με τη δικτατορία. Είμαστε όλοι πια αρκετά όριμοι για να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε τις εξουσίες της δημοκρατίας και να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι στεναρή η εδραίωση της δημοκρατίας της χώρας μας. Επομένως, όπως είπε στην προηγούμενη μου παρέμβαση, η νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία στην Αργεντινή προσπαθούν να εξασφαλίσουν το ότι θα υπάρχει διαλεύκανση της αλήθειας την εποχή της δικατορίας. Και προφανώς όλοι αυτοί που θέλουν να επισκεφθούν τη χώρα μου είναι καλόδεκτοι. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Ευχαριστώ τον δικαστή κύριο Ραφέκας ε, και τον δικηγόρο Γιανσόν. Ακούσαμε πολλές ιδέες για το πόσο στο μέλλον μπορούμε να δώσουμε σημασία στα όσα συμβαίνουν στην Αργεντινή και να τα υποστηρίξουμε. Και ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας ε, με, για τη σχέση με τις χώρες Μερκοσούρ τα άκουσε αυτά τα στοιχεία, άκουσε αυτές τις υποδείξεις. Και ελπίζω να έρθει σε επαφή και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δει τι άλλο μπορεί να γίνει. Επίσης, Υπάρχει μπροστά μας ένα μεγάλο καθήκον που πρέπει να προσπαθήσουμε να το προωθήσουμε, την διεθνή δικαιοσύνη και να δημιουργήσουμε, να βοηθήσουμε τις διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε την, ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είτε την ε, Αμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, δηλαδή είτε διεθνείς είναι οι οργανώσεις αυτές, είτε περιφερειακές, πρέπει να τις υποστηρίξουμε, ούτω ώστε οι ένοχοι όταν χρειάζεται Φερρυπίν να φτάνουν ενώπιον του Διεθνούς ε, ε, ποινικού δικαστηρίου. Ε, έχουμε πολλά αποθαρρυντικά στοιχεία, όπως με τον πρόεδρο του Σουδάν, Αλμπασίρ, ας πούμε, που δεν έφτασε ποτέ ενώπιον του Διεθνούς ποινικού δικαστηρίου. Ε, επίσης θα πρέπει να υπάρχει προστασία από την υποχρεωτική εξαφάνιση. Μετά από αυτά τα λόγια και αφού σας εκφράσω την ε, βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου που ήρθατε εδώ, νομίζω ότι υπάρχει και μια άλλη έκθεση που θα συζητήσουμε τους τελευταίους μήνες για τις α, μυστικές κρατήσεις. Ε, ο κύριος Νόβα και ο κύριος Σάινινγκ. Ο κύριος Σάινινγκ θα είναι παρόν, μας είπε. Ε, θα μιλήσουμε για αυτά τα κέντρα μυστικών κρατήσεων όπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε λαμβάνουν χώρα βασανιστήρια και φρικαλαιότητες. Όλα αυτά θα πρέπει να τα αποκαλύψουμε στα μάτια του κόσμου και θα πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη για τα θύματα. Αυτά σας ευχαριστώ. The Τέλειωσε η ακρόαση, αλλά όχι η συνεδρίαση. Καλωσορίζω την αντιπροσωπεία από το Βανουά του στην Επιτροπή μας. Ε, παρακολουθήσατε τις συζητήσεις. Είσαστε εδώ για την ε, συνέλευση ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας καλωσορίζω. Υπάρχουν αυτές οι ερωτήσεις τώρα των μελών ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Μπάρβαρα Λοχπίλερ έχει να κάνει κάποιε ερωτήσει, θα τι κάνει διαστόματο ε, κυρία Νίλσεν. Η Μπάρμπαρα δεν είναι εδώ. Θα ήθελα λοιπόν να διατυπώσω εγώ την ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την κατάσταση στη Ρουάντα είναι το ερώτημά τη. Ο πρόεδρος Πολ Καγκαμέ ε, έθεσε τέλος στη γενοκτονία τη Ρουάντα το 1994. Παρ' όλα αυτά η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρουάντα είναι ενισχυτική. Ε, στην λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό ε, μπαίνει ο στρατό, ε, ε κλίματα κατά αμάχων, δεν υπάρχει ελεύθερη αντιπολίτευση, ε, θύμωση του τύπου, δεν υπάρχει δυνατότητα τη ελεύθερη συνέβρεση ε, πολιτικές δολοφονίες. Πρόσφατα ο κύριος Ρουγκάν δημοσιογράφος δολοφονήθηκε, καθώς και ο εκπρόσωπος του Πράσινου Κόμματος, ο κύριος Ρουί Σερέκα, δολοφονήθηκε επίσης. Ε, το ερώτημα λοιπόν που θέλουμε να θέσουμε είναι αυτή η σιωπή της Ευρώπης για την κατάσταση των δικαιωμάτων στη Ρουάντα. Η Κομισιόν γνωρίζει την κατάσταση. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση πώς ερμηνεύει αυτά τα αιματηρά γεγονότα. Η Κομισιόν έχει έρθει σε επαφή με τις αρχές της Ρουάντας για να δοθούν διευκρινήσεις για τις εν λόγω δολοφονίες. Τι πληροφορίες έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκθεση που δεν δημοσιεύτηκε προς το παρόν, που γνωρίζουμε όλοι, γιατί διέρευσε στον τύπο για τα εγκλήματα των Ρουαντέζων στρατιωτών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονκό και για τις κατηγορίες αυτές περί γενοκτονίας. Τι έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Νίλσεν και τώρα έχει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιο θα απαντήσει από πλευρά Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Είμαι επικεφαλής της Μονάδας για την Κεντρική Αφρική. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία αυτή που έχω να απαντήσω. Είναι πολλά θέματα τα οποία τέτοισαν από την αξιότιμο κυρία Βουλευτή που έχουν να κάνουν με το τέλος της γενοκτονίας στην γενοκτονία μετά από το 1944 από τον πρόεδρο Καγάμε και την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με αυτήν. Ακολούθησε η κατάσταση που οδήγησε σε εκλογές στην Ρουάντα με επιθέσεις, με χειροβομβίδες, με δολοφονίες κτλ. Σε ό,τι αφορά την έκθεση του ΟΗΕ, το, το κείμενο αυτό που έχει διαρρεύσει στον τύπο είναι ένα, ακόμα ένα σχέδιο. Δεν είναι επίσημο έγγραφο. Ο στόχος μας είναι να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Μα ρωτούν αν η Κομισιόν γνωρίζει τα γεγονότα της Ρουάνδας. Μας λένε ότι τα ευρωπαϊκά όργανα έμειναν σιωπηλά και άπρακτα. Φυσικά είμαστε ενήμεροι, κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε στεναρά και ταχύτατα σε αυτά τα γεγονότα, στις δολοφονίες και τις ομότητες τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Έχω μαζί μου την δήλωση του εκπροσώπου, της υπάτου εκπροσώπου και αντιπροέδρου της Κομισιόν της κυρίας Άστον, η οποία ζητά να γίνουν οι απαραίτητες δικαστικές έρευνες και εξάλλου Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασιζόμενη στο άρθρο 8 της συνθήκης του Ισκοτονού στις 13 Ιουλίου και στις 8 Ιουνίου, ή Αυγούστου συγγνώμη, αντιμετώπισαν αυτό το θέμα. Η ερμήνεια της, των γεγονότων από την πλευρά της Κομισιόν ποια είναι. Κατά την άποψή μας, χωρίς να ξέρουμε ποιος βρίσκεται πίσω από αυτές τις δολοφονίες και τις χειροβοβικές επιθέσεις, θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι μια στρατηγική αποσταθεροποίηση στην Ρουάντα. Μέχρι στιγμή, βάσει των πληροφοριών μας, Συνεχίζονται οι δικαστικές ερεύνες στην περίπτωση του δημοσιογράφου Jean Leonard Rougambaki. Συνελήθησα τέσσερις μέρε μετά την, την επίθεση εναντίον του δύο υπόπτυο και ο σύμφωνα με τις έρευνες, ήταν το 1994 μέλος μιας ε, ομάδος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι υπήρξε μια αντεκδίκηση που οδήγησε στον φόνο του. Ο κύριος Διντάς, ένας από τους υπόπτους, βρίσκεται σε κράτηση και ο, κύριος, και ο δεύτερος ύποπτος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ελευθερία. Η δίκη τους που έπρεπε να γίνει 27 Σεπτεμβρίου γίνεται τώρα στις 8 Οκτωβρίου για να μπορούν να συμμετέχουν οι συνηγοροί τους. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Ανδρέ Καγουά, τη δολοφονία του. ένα ύποπτο συνελήφθη και αφέθη ελεύθερος τον Αύγουστο και συνεχίζουν οι έρευνε από την αστυνομία. Κυρία Πρόεδρε, η αντιπροσωπεία μας εξακολουθεί να παρακολουθεί τι περιπτώσει αυτέ, το των μάλλον καθώσεων, διότι ο πρόεδρος της ομάδας των Πρασίνων ζήτησε να γίνουν, του κόμματος των ζήτησε να βρεθούν οι ύποπτοι και να έλθουν ενώπιον της και ο άρθρο του 8, 8 της Συμφωνίας της Κοτονού θα χρησιμοποιηθεί από την πλευρά της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και είμαι στη διάθεση σα να απαντήσω σε περαιτέρω ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Κάγκαμε. Αώρα. Η κυρία Κιλ Νίλσεν, εξ ονόματος της κυρίας Ροκτουφάιλ. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Ας πάμε στην ερώτηση της κυρίας Κιλ Νίλσεν. Δική της ερώτηση. Είναι προσωπική δική μου ερώτηση που αφορά τον Κούρδων της Τουρκίας. Μια δίκης που θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της δίκης, 151 άτομα, μεταξύ, των, μεταξύ 1.500 Κούρδων που έχουν συλληφθεί εδώ και 18 άτομα, 151 λοιπόν άτομα, τρει παλιοί βουλευτές, 25 δήμαρχοι ή πρώην δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι θα δικαστούν. Ο κύριο Όσπαν Μπαϊντεμίρ, ο Δήμαρχο του Ντιέρ Μπακίρ, ε, μεγάλη πόλη, βασική πόλη του Κουρδιστάν, είναι ένα άτομο το οποίο γνωρίζω, γιατί ήμουνα αντιδήμαρχος της ε, ΡΕΝ που είχε συνεργασία με τον Ντιερμπακή το γνωρίζω τον Δήμαρχο, τον ε, υποδεχθήκαμε στη ΡΕΝ, ε, μας υποδέχθηκε εκείνος στην ε, πόλη του. Είναι αξιοσέβαστο άτομο και φιλιρινικός. δεν μπορεί λοιπόν από τον Ιανουάριο το τον περασμένο να φύγει από την Τουρκία, μαζί επίσης με τον αντιπρόεδρο της οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που είναι η μεγαλύτερη οργάνωση στο, των Κούρδων. Αυτός λοιπόν είναι φυλακισμένος εδώ και ένα χρόνο. Ε, Λέλα Γκιουβέν και Σεμούς Μπεϊάν επίσης, επίσης έχουν ε, συρθεί ενώπιον ενός δικαστηρίου. Διερωτώμε λοιπόν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι γίνεται με αυτές τις δίκες που έχουν ε, σαφώς πολιτικό χαρακτήρα. Τι πρωτοβουλίες έχουν αναλυθεί για να παρακολουθήσετε την κατάσταση των πολιτικών αυτών κρατουμένων. Η Τουρκία, η οποία σε καμία περίπτωση δεν πληρεί τα κριτήρια της Κοπενχάγης σε ό,τι αφορά το σεβασμό των μειονοτήτων. Τι γίνεται με τις συζητήσεις σας με την Τουρκία ε, για αυτά τα θέματα. Πώς μπορεί η Τουρκία να λάβει υπόψη και να σεβαστεί τις μειονότητες και τα, δικαιω... και τα δικαιώματά τους. Και επίσης, για τη δίκη της 18 η Οκτωβρίου, η Κομισιόν θα στείλει παρατηρητές. Αυτά είχα να ρωτήσω. Ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Ευχαριστώ, κύριε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κίλς Νίλσεν. Είμαι επικεφαλής μονάδος στην Γενική Διεύθυνση Διεύρυνση για την Τουρκία και επομένω υπεύθυνο για τα πολιτικά θέματα για την Τουρκία και τη διαδικασία διεύρυνση βάσει του προγράμματο το οποίο είχε καθοριστεί. Θα έπρεπε να ήμασταν στις 16.45 ο αρμόδιος χάρη στη θαυμάσια σας ε, Προεδρία κυρία Χάουταλα τα πράγματα έχουν επιταχυνθεί. Τρέχον είναι στο διάδρομο ο εκπρόσωπος τη Επιτροπής για τα θέματα αυτά. Ίσως θα πρέπει να επιτρέψει στον κύριο Ζων Κριστόφ Φιλορί να έρθει εδώ. Ίσως μπορούμε να περάσουμε στο θέμα τη Ρωσία και διεκπεραιώνουν τα επόμενα θέματα. Θα δώσω χρόνο στον κύριο Φιλορί για να απαντήσω στην κυρία Κίλς Νίλσεν. Η uh, Βλέπω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ότι συνέβη καταφατικά η κυρία Κίλς Νίλσεν. Θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Αντρικάινα να παρουσιάσει και το δικό της ερώτημα και ίσως θα επανέλθουμε στο ερώτημα της Νίλς Κίλσεν. Σας ευχαριστώ. Το ερώτημά μου αναφέρεται τις διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ξεκίνησαν πριν από πέντε χρόνια, το 2005, αυτές οι διαβουλεύσεις και μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το εξή ότι τα θέματα αυτών των διαβουλεύσεων περιλαμβάνουν την ε, κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία και το υπόλοιπο της, ε, του Βόρειου Καυκάσου περιλαμβάνοντας την κακομεταχείριση και τα βασανιστήρια. Το ερώτημά μου είναι ποια, ποιο είναι το περιεχόμενο αυτών των συζητήσεων στις επαφές Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Ποια είναι, η κατάσταση, θέση της Ρωσίας σε σχέση με τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία και στον υπόλοιπο Κάφκασο και τη Βόρεια Οσετία συγκεκριμένα. Τι έχει να πει η Ρωσία σε σχέση με τα τραγικά γεγονότα στο Μπεσλάν το 2004. Αν έχει συζητηθεί εξάλλου το θέμα αυτό ποτέ σε αυτές τι συζητήσει και τι συμβαίνει με τα δικαιώματα των συγγενών των φωνευτέντων στο Μπεσλάν, το δικαίωμά του για την πληροφόρησή του, για την επιχείρηση αυτή και την τύχη των θυμάτων και επίσης την ευκαιρία που έχουν να αναγνωρίσουν τους οικείους τους που υπήρξαν θύματα. Ποια ήταν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αυτών των διαβουλεύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ανδρίκενα. Για τους μη γνωρίζοντες, η κυρία Ανδρίκενα και εγώ και ο κύριος Μπέρμαν επισκεφθήκαμε το σχολείο στο Μπέσλαν όπου είδα τα τραγικά γεγονότα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Χαουτάλα και ευχαριστώ και την κυρία Ενέ για την ερώτηση, η οποία είναι και επίκαιρη. Γιατί πρόσφατα ήταν η επέτειος των δολοφονιών στο σχολείο Μπέσλαν, το Σεπτέμβριο δηλαδή. Κυρία Αντρικίνε, θέλω να σα διαβεβαιώσω ότι η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βόρειο Κάφκασο και στην Τετσενία όλο ιδιαίτερο. ιδιαίτερος ε, με όλα τα ζητήματα που θέσατε ε, είναι στην ατζέντα των διαβουλεύσεων που έχουμε τη Ρωσία το 2005 για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα μπορούσα να πω και κάτι παραπάνω μάλλον, μάλιστα, ε, να σας πω ότι η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βόρειο Κάφκασο είναι κεντρικό σημείο των συζητήσεών μας από το 2005 των διαβουλεύσεων αυτών. Στην πρόσφατη, τελευταία συνάντηση που είχαμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά επανάληψη έκανε έκκληση στη Ρωσία να εισάγει συγκεκριμένα μέτρα για να αντιμετωπίσει την ατιμορρησία ειδικά στον, τομέα των διοκτικών αρχών. Έχουμε εκφράσει ανησυχίε για την ε, δύσκολη κατάσταση. Δύσκολη είναι φημισμό σε ό,τι αφορά την κατάσταση των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι πρέπει να την προστατεύσουμε. Επίση, έχουμε τονίσει τη σημασία τη απόδοση δικαιοσύνη προ τα θύματα και ενθαρρύνουμε στεναρά τη Ρωσία για να βελτιώσει το διάλογο με την κοινωνία των πολιτών ε, σε όλο το Βόρειο Κάφκασο, όπου η κατάσταση εξακολουθεί να επιδεινώνεται. Τώρα, ποια ήταν η απάντηση της Ρωσίας σε όλα αυτά, στις συζητήσεις Οι Ρώσοι μας έδωσαν απαντήσεις σε μεμονωμένες περιπτώσεις που τονίσαμε και θίξαμε. Οι Ρώσοι αναγνώρισαν ότι η κατάσταση ασφαλείας στο Βόρειο Κάφκασο έχει επιδεινωθεί περαιτέρω. Και αναγνώρισε ότι η κατάσταση των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει επιδεινωθεί αυτό δεν διαφεύγει, δεν διέλαθε της προσοχή των πολιτικών ηγετών της Ρωσίας. Ε, γνωρίζουν τις δολοφονίες ε, των υπερασπιστών και ακτιβιστών α, των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Το γνωρίζει και ο πρόεδρος και ο γενικό γενικός εισαγγελέας. Ο πρόεδρος Μεντέντεφ έχει μια στρατηγική σε πέντε σημεία για να καταπολεμήσει την τρομοκρατία στο Βόρειο Κάφκασο και είναι κάτι που συζητήσαμε πολύ στις τελευταίες μας επαφές. Η ευρωπαϊκή πλευρά καλωσορίζει τη σφαιρική προσέγγιση του Προέδρου, αλλά κάναμε έκκληση στη, πλευρά να προωθήσει συστηματικές μεταρρυθμίσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τις δολοφονίες του 2004 στο σχολείο αυτό, αυτό το θέμα ε, το είχαμε συζητήσει στις προηγούμενες επαφές ε, που είχαμε το 2005 και 2006 ε, και κατά επανάληψη συζητήσαμε την αποζημίωση προς ε, τα θύματα των επιχειρήσεων αντικτρομοκρατίας. Επίσης, κρατάμε αυτό το διάλογο ανοιχτό μέσω του καναλιού της ΟΑΣΕ. Τον Νοέμβριο θα έχουμε την επόμενη διαβούλευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη Ρωσία και μην ξεχνάτε ότι πάλι ο Βόρειος Κάφκασος θα είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί από τα πρώτα. Θα συζητηθεί διεξοδικά του κράτου δικαίου, ε, της κοινωνία των πολιτών, της δικαιοσύνης, ε, την κατάσταση των ε, γυναικών επίσης στην περιοχή. Αυτά θα είναι τα πιο συγκεκριμένα θέματα που θα συζητήσουμε σε επαφές μας τον Νοέμβριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπω είπε η Χάιντι Χάουταλα, ήμασταν στο Μπεσλάν στι αρχέ του Σεπτεμβρίου, στην Βόρεια Οσετία και, στο, και στην Ιγκουσιωτία. Και είχαμε επαφέ με τι μητέρε και του οικείου των θυμάτων στο σχολείο στο Μπεσλάν. όπω ξέρετε έγιναν πριν από 6 χρόνια αυτά τα τραγικά γεγονότα. Αυτό το οποίο μάθαμε εκεί είναι ότι συνεχίζονται ακόμα οι έρευνε για το τι ακριβώ συνέβη και δεν έχουν πρόσβαση εκεί των θυμάτων στις πληροφορίες αυτές που προκύπτουν από τις έρευνες του ζητήθηκαν να αναγνωρίσουν σώματα, ζήτησαν να αναγνωρίσουν τα, τα λείψανα των οικείων τους που βρίσκονται θαμένα στο νεκροταφείο τους αρνήθηκαν αυτό το δικαίωμα. Επίσης, στον Εσραν, στην Ιγκουσετία, συναντήσαμε άτομα τα οποία είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι εκεί. Πρόκειται για άτομα τα οποία πριν από 18 χρόνια εκδιώχθηκαν από τις αιστείες τους, από το έδαφος που είναι τώρα η Βόρεια Οσετία εκδιώχθηκαν στην Ιγκουσετία. Τα άτομα αυτά, και είναι χιλιάδες, 25.000, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, και δεν έχουν κανένα νομικό καθεστώς. Δεν έχουν καμία δυνατότητα να ζητήσουν κοινωνικές παροχές. Και ακούσαμε ανατριχιαστικές ιστορίες από όλα αυτά τα άτομα. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το, μάλλον η αίτησή μου είναι να τεθεί αυτό το θέμα στα πλαίσια του διαλόγου ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη Ρωσία, γιατί η Ρωσία είναι και στρατηγικός μας εταίρος. Και η στρατηγική μας ε, σχέση πρέπει να βασίζεται σε αξίες και τα ανθρώπινα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε Αντρίκενα. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει να πει κάτι. Πάρα πολύ σύντομα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πραγματικά για αυτή τη μαρτυρία, για όσα είδατε εκεί εσείς δύο σώμασοι. Είναι πάρα πολύ καλό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχουν τέτοιε μαρτυρίε και βέβαια το δεύτερο είναι φυσικά θα παρακολουθήσουμε και θα δώσουμε συνέχεια και με τους συναδέλφους που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και πάντα να θέτουμε υπόψη τους αυτά τα θέματα ακριβώς και επειδή είμαστε σε επαφή μαζί σας. Όταν συζητούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την ευκαιρία να προβάλλουμε και εμείς και να ε, αντιπροσωπεύουμε τι τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, θα έρθω σε επαφή με τους συναδελφούς που ασχολούνται με αυτό το θέμα και κάνουν αυτό το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να δούμε τι μπορεί να μπει στην μέση διάταξη Γνωρίζω και δυστυχώς ότι ο Βόρειος Κάφκασος είναι πάγιο θέμα στη Μέση Διάταξη λόγω της καταστάσεως εκεί. Δυστυχώς ελπίζω κάποια στιγμή να βγει γιατί θα έχουν βελτιωθεί τα πράγματα αλλά προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται. Ευχαριστώ κύριε Χέρτς. Είμαι βέβαια, βέβαια ότι από κοινού θα μπορέσουμε να προτείνουμε κάποιες λύσεις για την περιοχή. Ενισχύουμε πάρα πολύ όταν συζητούμε ιδίω με τα θύματα και τους συγγενείς των θυμάτων που έχουν δολοφονηθεί, εξαφανιστεί και τα λοιπά και βασανιστεί. Τελευταία ερώτηση δική μου για τη Ρωσία. Είναι γνωστή η περίπτωση του δικηγόρου Σεργέη Μπαγνίτσχη που ήταν προφυλακισμένος και έχασε τη ζωή του στη φυλακή στη Μόσχα στην ηλικία των 37 ετών στις 16 Νοεμβρίου 2009. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι διώχθηκε γιατί ήταν ανένδοτος ο αγώνας του κατά της ε, απάτης και της διαφθοράς. Συνελήφθη από τους ίδιους αξιωματούχους τους οποίους κατηγορούσε για διαφθορά και μάλιστα πολύ μεγάλη κλίμακα ε, υπεξαίρεσης ε, εσόδων φορολογικών του ρωσικού κράτους από τους υπαλλήλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς κρίνει την αποτελεσματικότητα και την αμεροληψία της έρευνας που γίνεται και της ποινικής δίωξης του κυρίου Σεργέη Μαγνίσκη. Ξέρω ότι αυτό ετέθη η υπόψη του στο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ικανοποιημένη από την απάντηση και από την πορεία της δίωξης και αν όχι τι προτίθεται να κάνει. Γιατί από ό,τι φαίνεται είναι και ε, καταφανής και πάρα πολύ καλά τεκμηριωμένη η αστυνομική ε, ε, βία και νοφία. Ευχαριστώ. Είναι τραγικός ο θάνατος του κ. Μεντέσκη, ενώ ήταν προφυλακισμένος. Είναι κάτι το οποίο έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. παρακολουθήσαμε κοντά το θέμα αυτό και ξέρουμε ότι δεν υπήρξε κάποια σημαντική πρόοδος τη ε, έρευνα για τον θάνατο του ελόγου ατόμου μέχρι τώρα. Για μας παραμένει πάρα πολύ σημαντικό όλες οι καταγγελίες παραβίασης ανθρωπινών δικαιωμάτων στη Ρωσία να τύχουν πλήρους και αποτελεσματικής έρευνας και οι δράστες τέτοιων αδικημάτων να έλθουν ενώπιον της δικαιοσύνης και έχουμε καταγράψει απόλυτα και έχουμε ε, καλωσορίσει την ε, δήλωση του κ. Μεντεβέντεφ ότι θα γίνει πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου κυρίου Μεντέσκη, Μανίσκη. Δυστυχώ δεν είναι μεμονωμένο γεγονό ο θάνατο του κ. Μανίσκη. Θα πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο μια συνολική κατάσταση και πάλι μπορώ να χρησιμοποιήσω τα λόγια του πρόεδρου Μεντεβέντεφ ότι υπάρχει ένα είδος δικαστικού μηδενισμού στην Ρωσική Ομοσπονδία Μέσα στα πλαίσια λοιπόν των επαφών που έχουμε με ε, τις ρωσικές αρχές ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθούμε να πιέζουμε για να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στις δικαστικές πρακτικές στην ε, Ρωσία και να υπάρξουν αποτελεσματικές έρευνες για καταγγελόμενες παραβιάσεις στο δικαστικό σύστημα και εξακολουθούμε να υπογραμμίζουμε το κατεπήγον του να υπάρξουν ουσιαστικές εκβάθρου μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα της Ρωσίας. Ο θάνατος κ. Μαγνίσκιτς μας γνίσκει μάλλον, οδήγησε σε κάποιες δράσεις από τον πρόεδρο Μετβέντεφ που θεωρούμε ότι είναι πολύ θετικές μέσα στα πλαίσια της ατζέντα εξυγχρονισμού στη Ρωσία. Μετά από τον, ε, τον τραγικό θάνατο του κ. Μαζνίσκη, ξεκίνησε ο πρόεδρος Μετβέντεφ μια μεταρρύθμιση στο, στο σύστημα των σοφανιστικών καταστημάτων, τροποποίηση του ποινικού κώδικου ώστε να μην υπάρχουν φυλακίσει σε τέτοιε περιπτώσει του κ. Μεσνίσκη και ε, μια σειρά νομοθετικών μέτρων ελήφθησαν που οδήγησαν στη θετική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπάτη εκπρόσωπος κυρία Άστον ήρθε σε επαφή και με τον κύριο ε, Μετβέντεφ και με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Λαύροφ για τα θέματα του κράτους δικαίου στη Ρωσία και όπως είπα προηγουμένως θα έχουμε Στι 17 Νοεμβρίου την επόμενη συνάντηση για διαβούλευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη Ρωσία και θα θέσουμε και πάλι το θέμα του κράτου δικαίου και τη δικαστική εξουσία και τα αυτά είναι μόνιμα θέματα στις συζητήσεις μα με τη Ρωσία και είναι πάντα στην κορυφή τη ημερησίας διαταξή μα. Πάλι στις 17 Νοεμβρίου θα τα θίξουμε με τη Ρωσία. Προσβλέπουμε λοιπόν στο να αντιμετωπίσουμε και μονομένε περιπτώσεις όπως αυτή του κ. Μιτβέτσικη. Παραδεχόμαστε επίση ότι παρά την ρητορική του κ παρά την συνέχιση της διεθνούς και εσωτερικής πίεσης στη Ρουσία, μέχρι στιγμής δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία κατά μηδενός σε σχέση με αυτή την περίπτωση, ούτε έχουν γίνει περαιτέρω έρευνες σε σχέση με την περίπτωση διαφθοράς στην οποία ο κ. εργαζόταν πριν από τον θάνατό του. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο, το, το Μάιο 2010 σε μια συνάντηση στο Καζάν εξέφρασαν τις σοβαρές ε, ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά στους ομολόγους, τους υπουργούς εσωτερικών. Μέχρι στιγμής η περίπτωση Μαγνίσκη παραμένει λιδία λίθος του αν ο πρόεδρος Μετβέντεφ είναι πράγματι προσιλωμένο σε μια μεταρρύθμιση στη Ρωσία και στο πνεύμα αυτό θα εξακολουθήσουμε να τονίζουμε τη σημασία αυτής της περιπτώσεως και άλλων παρομοίων περιπτώσεων στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σε όλες τις επαφές μας με τη Ρωσία. Ευχαριστώ. Με μεγάλη χαρά άκουσα ότι θα συνεχίσετε να διερευνάτε το θάνατο του κ. Μαγνίσκης. Αναγνωρίζετε και εσείς δεν υπάρχουν αποτελέσματα μέχρι στιγμής, παρά την προσπάθεια του Προέδρου για να γίνει μια πραγματική διερεύνηση των αιτίων θανάτου. Αλλά όπως είπατε και εσείς δεν είναι μεμονωμένο αυτό το περιστατικό. Στις διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εταίροι μα στις συζητήσεις είναι κυρίως η εταίρη σας μάλλον, είναι το Υπουργείο Εξωτερικών. Και από ό,τι κατάλαβα και εγώ και στην αδελφή μου που παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα, καλό θα ήταν και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών να έρθουν και αυτοί στο, στην τράπεζα των συζητήσεων για να συζητήσουν για, για τις μεταρρυθμίσεις του σοφωνιστικού συστήματος και τις παραβιάσεις και υπερβάσεις και καταχρήσεις αρμοδιοτήτων της δικαιοσύνης. Θα ζητήσετε λοιπόν και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών να εμπλακούν στις διαβουλεύσεις αυτές. Ευχαριστώ κυρία Χαουτάλα. Σωστή ερώτηση. Το 2005 απογοητευθήκαμε με τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και τη στάση των Ρώσων, οι οποίοι αντιμετώπισαν τις ε, διαβουλεύσεις αυτές ως ενδιαφέρουσες κτλ. Αλλά καθαρά σε διπλωματικό επίπεδο. Όπως και με την Κίνα, υπάρχει και με τη Ρωσία μια διαδικασία διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ακριβώς ένα από τα σημεία για τη μεταρρύθμιση του διαλόγου είναι αυτό το σημείο που θέσατε. Φυσικά η, η κυρία Άστον όταν Μάλστρομ, όταν συναντηθεί με τους ομολόγους της από το, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, καλό θα ήταν να θέσει και αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ. την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις απαντήσεις της. Στο τέλος των ερωτήσεων μας έχουμε φτάσει. και θέλω να χαιρετήσω και την παρουσία. Α, συγγνώμη, ο κύριος Φιλωρή έχει έρθει. Ο εμπειρογνώμων της Τουρκίας έχει έρθει. Ο κύριος Φιλωρή είναι μαζί μας. Βεβαίω, συγγνώμη κύριε Φιλωρή. Νομίζω ότι γνωρίζετε πλέον το ερώτημα, οπότε μπορείτε να απαντήσετε αν θέλετε. Κύριε Φιλωρή, έχετε το λόγο. Ναι, ναι. Έχει έρθει η Τουρκία, κυρία Χάουταλα, πράγματι. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά υποδεχόμουνα εκπροσώπους της Τουρκίας που μου θέτανε ορισμένα ζητήματα για την ελευθερία έκφρασης και ελευθερία τύπου στην Τουρκία. Για το συγκεκριμένο σας ερώτημα. Η Κομισιόν παρακολουθεί από κοντά την υπόθεση αυτή που οδήγησε στην απαγγελία κατηγορία εναντίον 150 ατόμων με την κατηγορία της υποτιθέμενης συμμετοχής τους στην πολιτική πτέρυγα του PKK γνωστή ως του PKK Κόγκραγκέλ, που είναι γνωστή ως KCK στα τουρκικά. Η απαγγελία αυτή καταγορίας έγινε δεκτή από τα δικαστήρια τον Ιούνιο του 2010. Η πρώτη ακρόαση σε δικαστικό επίπεδο θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου του 2010 στο ε, δικαστήριο στο Κακούργιο Δικείο του Διαρμπακύρ. Στις 12 Νοεμβρίου προβλέπεται να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία και θεωρώ ότι λόγω της σημασίας αυτού του προβλήματος θα υπάρχουν εκατοντάδες ουσιαστικά δικηγόροι οι οποίοι θα λάβουν το λόγο κατά τη διάρκεια της δίκης. Οι περισσότεροι κατηγορούμενοι, 104 συνολικά, παραμένουν στην φυλακή αναμένοντας την ε, δίκη τους και οι άλλοι 47 ε, ακόμα 47 κρατούμενοι είναι ελεύθεροι. Γνωρίζει η Κομισιόν ότι ο κ. Μουχαρέμ Ερμπέι ε, αντιπρόεδρος της ε, Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων IHD και πρόεδρος του κλαδικού τμήματος στο Diyarbakir της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένας από αυτούς οι οποίοι είναι υπόδικοι αυτή τη στιγμή. Και βάσει των πληροφοριών που έχουμε ο κύριος Ερμπέι κρατείται στις φυλακές τύπου D του Διάρμπακ αναμένοντας την δίκη του οι υπηρεσίε της Κομισιόν έχουν θέσει το θέμα αυτό του κυρίου Ερμπέη ενώπιον των τουρκικών αρχών κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης για τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεχάης στις 15 Απριλίου 2010 στην Άγκυρα και πρέπει μπορώ να σας επιβεβαιώσω επίσης ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Άγκυρα θα είναι παρόν στις 18 Οκτωβρίου στην πρώτη δικαστική στην πρώτη ακρόαση στα δικαστήρια, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία και την βαρύτητα των κατηγοριών εναντίον των κατηγορουμένων, η Κομισιόν προσδοκά ότι η διαδικασία αυτή θα γίνει με πρέποντα σεβασμό των κανόνων δικαίων και με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων. Σε πιο γενικό επίπεδο θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω το ότι, παρά το γεγονός ότι η Κομισιόν έχει απόλυτη αλληλεγγύη με τον τουρκικό λαό στον αγώνα του κατά της τρομοκρατίας θεωρεί επίσης ότι τα μέτρα αντιτρομοκρατικού χαρακτήρα δεν θα πρέπει να γίνονται σε βάρος των βασικών δημοκρατικών ελευθεριών. Είχαμε εν καιρό χαιρετήσει τη δέσμευση της τουρκικής κυβέρνηση στη λεγόμενη δημοκρατική, στο δημοκρατικό άνοιγμα για την αντιμετώπιση και του κουρδικού θέματος. Όλα αυτά τώρα πρέπει να αναζωογονηθούν για να μπορέσουν να καλύψουν τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν εκείνη την εποχή. Καταγράψαμε με ικανοποίηση ότι το τουρκικό κοινοβούλιο τον Ιούλιο, η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, τροποποίησε την νομοθεσία η οποία αφορά ανήλικους παιδιά τα οποία ε, διαπράττουν αδικήματα και πια προβλέπεται να δικάζονται σε δικαστήρια ανηλίκων. Διότι θυμόστε, θυμόστε στο παρελθόν τα παιδιά αυτά τα οποία κατηγορούνται για εγκλήματα τρομοκρατικού χαρακτήρα ε, έρχονται ενώπιον ποινικών δικαστηρίων για ενηλίκους, κάτι το οποίο απασχόλησε ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα θα αντιμετωπίζονται από ειδικά δικαστήρια ανηλίκων και μόνο. Οι προσπάθειες για να βελτιωθεί η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην νοτιοανατολική Τουρκία θα πρέπει να συνεχιστούν. Καταγράφουμε με ανησυχία σχετικά την αύξηση σε πιέσει κατά των εφημερίδων που συζητούν τα κουρδικά θέματα ή δημοσιεύουν άρθρα στα κουρδικά. Επίση, οι διαδηλώσει στο νοτιοανατολικό τμήμα τη ε, Τουρκία σε σχέση με το κουρδικό θέμα εξακολουθούν να σημαδεύονται από βία γεγονότα. Έχουμε κατ' επανάληψη τονίσει σε πολλέ ευκαιρίε και το λέμε και τώρα πάλι και το έχουμε πράξει φυσικά αυτό και στι εκθέσει πρόοδου μα σε σχέση με την Τουρκία, ότι θεωρούμε ότι η αντιτρομοκρατική νομοθεσία στην Τουρκία θα πρέπει να τροποποιηθεί για να αποφευχθεί μια υπερβολικά διασταλτική ερμηνεία αυτη τη νομοθεσια που έχει οδηγήσει σε ένα δυσανάλογο υψηλό άτομο κρατουμένων οι οποίοι συνδέονται με υποτιθέμενες τρομοκρατικε πραξει Και πάλι θα κάνουμε μια έκθεση για την πρόοδο τη Τουρκία προ την επίτευξη των κριτηρίων Κοπεχάγης για προσχώρηση στην επόμενη έκθεση πρόοδου η οποία θα προβλέπεται να δημοσιευτεί στις 9 Νοεμβρίου. Η ανάλυση μας θα βασιστεί σε μια ισοδίκαια και πραγματική ανάλυση δεδομένων που θα έλκονται από διάφορες πηγές μεταξύ των οποίων και μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ανατολικό τμήμα της Τουρκίας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Κιλ Νίλσεν έμεινε ικανοποιημένη από την απάντηση. Προς το παρόν ναι και προτίθεμαι και εγώ από πλευρά μου να παρακολουθώ πολύ κοντά αυτή την υπόθεση. Ωραία. Τώρα μπορούμε να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις απαντήσεις που μας έδωσε και βεβαίω θα παρακολουθούμε αυτά τα θέματα και στο μέλλον. Και ένα τελευταίο τώρα. Θα ήθελα να καλέσω δύο εξέχοντες ε, ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Σουδάν στην Επιτροπή να τους καλωσορίσω. Χάνια Καβά, που ήταν επικεφαλής ε, ενός ε, κέντρου στην Χαρτούμ και συντόνισε την εκστρατεία ε, προσυπογραφής και κύρωσης της σύμβασης κατά των βασανιστήριων και άλλων απάνθρωπων πρακτικών. Χρειάστηκε να φύγει από τη χώρα του γιατί διωκόταν ε, αυτή τη στιγμή εκδόθηκε ε, ασκήθηκε μάλλον δίωξη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Πρόεδρου Αλμπασίρ και ε, δίπλα του κάθεται ο κύριος Αμπτελμόνιμ Ιμπκακ που είναι γνωστός δικηγόρος για την καταπολέμηση της ατιμορρησίας στη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα συνελήφθη στη δεκαετία του 90 μετά το πραξικόπημα που έφερε την τωρινή κυβέρνηση στην εξουσία. Ε, συνελήφθη στη Χαρτούμ στις 24 Νοεμβρίου στη συνέχεια του 2008 μαζί με δύο συναδέλφους υπέστη βασανιστήρια και άλλες ε, κακοποιήσεις κατά τη διάρκεια της φυλαξή του. Στη συνέχεια μόλις αφέθηκε ελεύθερος έφυγε ε, και κυρίως τρέφει ε, στην Καμπάλα και στην Τζούμπα το Δεκέμβριο του 2009 κατέθεσε μήνυση κατά των αρχών του Σουδάν για τη μεταχείριση ε, που είχε υποστεί τον Νοέμβριο του 2008. Μήπως θέλετε να λάβετε το λόγο για λίγα λεπτά, να εξηγήσετε ποια είναι τα βασικά προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν αυτή τη στιγμή um, και να μας πείτε αν είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε με την κυρία Ρόζα Λίντ Μάρστεν που είναι η ε, νέα ε, ύπατη πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί και ήταν χτες στην ε, Επιτροπή Εξωτερικών. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θέλω σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να μεταφέρω τις ανησυχίες των αγωνιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Σουδάν σε αυτήν την δύσκολη στιγμή που διατρέχει το Σουδάν. Σε 100 μέρες περίπου ο λαός του Νότιου Σουδάν θα κληθεί σε δημοψήφισμα για να εκφράσει το δικαίωμά του για αυτοδιάθεση. Ένα ειρηνικό δημοψήφισμα θα λάβει η χώρα στις 9 Ιανουαρίου, κάτι το οποίο δεν, ήταν, δεν θα ήταν δυνατόν να λάβει χώρα όσο η κυβέρνηση εξακολουθεί να υπονομεύει και να υποσκάπτει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Σουδάν. Το δικαίωμα αυτοδιάθεσης και η αναγνώριση του αποτελέσματος είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να εμποδιστεί η έκρηξη βιαίων γεγονότων όπως φοβούνται πάρα πολύ οι εκλογές του προηγούμενου Απριλίου με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας δεν συνοδεύτηκε από την απαραίτητη μέρημνα για την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων μεταξύ των οποίων το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε και το δικαίωμα του έκφρασης που είναι απαραίτητα για την ιδευρέωση των πολιτικών δικαιωμάτων στη χώρα μας. Μετά από τις εκλογές αυτές οι εθνικές μυστικές υπηρεσίες έδρασαν και σώβησαν κατά των μέσων ενημέρωσης, των αγωνιστών κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων και των αντιφρονούντων όλων αυτών λοιπόν οι οποίοι υποστήριξαν την ελευθερία του τύπου βρέθηκαν σε καταδίωξη. Χρειάζεται η υποστήριξη λοιπόν όλων αυτών των αγωνιστών που αγωνίζονται για μια ελεύθερη κοινωνία και ελεύθερα μέσα ενημέρωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ζητήσει να υπάρξει διεύρυνση τη εντολή του, ανεγνω... του ανεξάρτητου εμπειρογνώμου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Σουδάν. Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίσει την εφαρμογή των κατευθυντηρών γραμμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των αντιφρονούντων και αγωνιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Σουδάν ώστε να μπορέσει να υπάρξει πλήρης ελευθερία για τα θέματα αυτά στην χώρα αυτή. Μετά από 7 χρόνια εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε μια ανθρωπιστική κρίση στο Ντάρφουρ η οποία σε μεγάλο βαθμό δημιουργήθηκε από την κεντρική κυβέρνηση στο Ντάρφουρ. Η στρατηγική για το Ντάρφουρ που έχει παρουσιαστεί εξακολουθεί να μην περιλαμβάνει και την ε, προστασία της, ε, των πολιτικών δικαιωμάτων, την ειρήνη και την ε, εδραίωση του κράτους δικαίου. Είναι μια... Το θέμα των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να ληφθεί υπόψη από οποιαδήποτε μορφή παρέμβασης στην περιοχή αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εξακολουθούμε να σας υποστηρίζουμε. Η κυρία Γκόμες έχει το λόγο, γνωρίζει τα τεκτενόμενα στο Σουδάν. Υποστηρίζω και συμφωνώ με τα όσα είπε ο φίλος μας από το Σουδάν. Έχω πάει στο Σουδάν πρόσφατα, στη διάρκεια των εκλογών και μία από τις συστάσεις μας προς το Κοινοβούλιο ήταν να δοθεί προσοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη όλους όσους ε, υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Σουδάν, στο Χαρτούμ και αλλού. Αυτή η σύσταση προέκυψε από την αίσθηση που υπάρχει ότι δίδεται υπερβολικά πολύ προσοχή και προτεραιότητα στο θέμα του δημοψηφίσματος στο Νότιο Σουδάν και ότι αγνοούμε τη μάχη των ανθρώπων υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν. Γι' αυτό λοιπόν είμαι εντυπωσιασμένη από την ζωτικότητα της, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Ο κύριος Σαλή Μαχμούτο Σαν Οσμάν πήρε το βραβείο Ζαχάροφ, Σουδανός, και η κοινωνία των πολιτών στο Σουδάν και στο Βόρειο Σουδάν ε, όλος ιδιαίτερος ε, αξίζει και αυτή της προσοχής μας. Δεν πρέπει να δώσουμε προσοχή μόνο στο δημοψήφισμα στο Νότιο Σουδάν και να γνωρίσουμε όλα τα υπόλοιπα θέματα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για το Σουδάν, ε, για το λαό του Σουδάν, είτε βρίσκεται στο βορρά είτε στο νότο η διαδικασία εκδημοκρατισμού στο Βόρειο Σουδάν είναι πολύ σημαντική. Επίσης, συμφωνώ με την άποψη ότι δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια προς στα όσα συμβαίνουν στον Ταρφούρ. Νομίζω ότι αδιαφορούμε για τον Ταρφούρ, πρέπει να, το, να δώσουμε σημασία στο τι συμβαίνει εκεί και θα πρέπει το Κοινοβούλιο να πιέσει τις αρχές, να κάνει κάτι πέρα από τα λόγια. Καλά είναι και τα λόγια, ειδικά της είπα της εκπροσώπου της κυρίας Άστον πριν από λίγες εβδομάδες ε, προς τις αρχές της Κένιας που δεν συνέλαβαν τον πρόεδρο Αλμπασίρ με βάση το ένταλμα που είχε εκδοθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αυτό είναι σημαντικό θέμα. Θα πρέπει οπουδήποτε, όποτε συζητάμε με τους Αφρικανούς φίλους μας, στα πλαίσια της ΑΚΕ, στα πλαίσια της Αφρικανικής Ένωσης, να το θέτουμε. Νομίζω ότι οι ευρωπαϊκές αρχές έδειξαν μεγάλη αδυναμία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκόμους. Κάθε επιτυχία στο σημαντικό σας έργο. Θα παρακολουθήσουμε αυτό το οποίο κάνετε και η νέα ύπατος η δική μάλλον εκπρόσωπό μα θα δώσει μεγάλη σημασία στην τοπική πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπείας στο Χαρτούμ. Θα είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπάρξει υποστήριξη στου αγωνιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα σα και εκτό αυτή. Ευχαριστώ. Και τώρα καταγράφουμε την επόμενη συνεδρίασή μας. Θα λάβει η χώρα την επόμενη Τρίτη στι 5 Οκτωβρίου, 3 η ώρα το απόγευμα μέχρι τι 4.30 είναι η δική μα κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων αλλά και με την Επιτροπή Ανάπτυξη για να ακούσουμε παρατηρήσει, παρουσιάσει μάλλον, για τι εννέα προτάσει για το βραφείο Σαχάροφ 2010. Μέχρι την επόμενη Τρίτη και η επόμενη συνεδρίασή μα, τακτική συνεδρίαση, θα γίνει στι 14 Οκτωβρίου, αν το θέλει ο Θεό, στι 9 το πρωί. Σα ευχαριστώ πολύ. Κλείνω τη συνεδρίαση.